Members, ε, καλημέρα. Ας ε, ξεκινήσουμε τους μαραθώνιους ψηφοφοριών. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τη συνάντηση των συντονιστών εχθές το βράδυ όσον αφορά τη ΣΟΑ. Είχαμε δύο θέματα. Πρώτον, ε, πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει τις ε, δυνατότητες ε, οδηγήσεως και η κυρία Τίκαου και η κυρία Κουαντιάνα ολοκλήρωσαν το θέμα αυτό σε συνεργασία με τη Γραμματεία. Η Γραμματεία ζήτησε επίσης να παρουσιάσουμε μία ενημέρωση των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη ΣΤΟΑ για να γνωρίσουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι ε, συνεχίζεται ακόμη και είναι εν εξελίξη. Όσον αφορά τους εισηγητές και τους συντάκτες, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΑΚΕΟ ε, είναι ένα θέμα όπου αποφάσισαν οι συντονιστές να αναλάβει ο πρόεδρος ή ένας αντιπρόεδρος και όσον αφορά ο Γαλιλαίο και GPS οι συντονιστές ε, αποφάσισαν ότι η ΙΤΡΕ ή άλλως ε, είναι η ε, επικεφαλής επιτροπή και αυτοί θα αποφασίσουν. Όσον αφορά τις ε, μεταφορές αποφασίστηκε ε, ε, το χώρο μεταφορών αποφασίστηκε ότι το ΕΛΚ θα αποφασίσει για το συντονιστή το, επίσης όσον αφορά το θέμα των γενικών μεταφορών αποφασίσαμε να μην υπάρξει κίνηση η ECR ανέλαβε στο επόμενο θέμα την ε, ε, την ε, συζήτηση και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε σχετικά να μην κάνουμε καμία κίνηση όσον αφορά την, ε, ε, την οικονομία χαμηλό διοξιδίου του άνθρακος, ε, το ίδιο και για την εξοικονόμηση πετρελαίου και το ίδιο για τις μεταφορές γύρω από το μεσογειακό χώρο. Όσον αφορά την ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αναθεωρηθούν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει, θα προχωρήσει σε μία ανακοίνωση και θα γίνει μία γνωμοδότηση σύμφωνα με το σύστημα περιφοράς. Επίσης ε, είχαμε και κλεισμένων των θυρών μία συνεδρίαση για την μαύρη λίστα της τις αεροπορίες και για την επιτροπολογία ανέφερα ότι έχουμε εβδομαδιαίο ε, μια εβδομαδιαία εφημερίδα και όσον αφορά τον διάλογο βάσει των προτεραιοτήτων που μας έχουν καταρτήσει οι πολιτικές ομάδες εγώ υπέβαλα μία πρόταση που αναφέρεται στις έξι προτεραιότητες για το 2012 με κάποια μικρή αλλαγή και υπήρξαν και οι προτεραιότητες <clears throat> οι οποίες προσέθεσαν ένα έβδομο θέμα αλλά θα δούμε αν καταφέρουμε και καλύψουμε τις πρώτες έξι θα δούμε τι θα επιλέξουμε για έβδομη. Όσον αφορά τα άλλα θέματα για τη μεταφορά των ζώων, η προφορική ερώτηση για τη μεταφορά των ε, ζώων θα αναλυφθεί από την ε, ε, Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος αλλά μπορούμε να κάνουμε μια προφορική ερώτηση είναι θέμα στη διάκριση των πολιτικών ομάδων και αυτές θα αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν στο θέμα αυτό. Όσον αφορά την πρόσκληση για το Eurocontrol στο Μαστρίχτ. Ε, ο κύριος Γκρός επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να γίνει αυτή η επισκέψη στα πλαίσια της επισκέψεως στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη Γερμανία τον Ιούνιο. Ε, συνάντηση με τον Επίτροπο Κάλλας. Συμφωνήσαμε να στείλουμε μία επιστροφή στους Επιτρόπους Κάλλας και Χάν για ε, το θέμα του, οδικού συστήματος της Πολωνίας και ε, μία επιστροφή στον κύριο Κάλλας σχετικά με τις ε, με τα τέλη που επιβάλλονται εις τους επιβάτες. Όσον αφορά την αναθεώρηση του πράσινου πακέτου, ε, για τους σιδηροδρόμους αποφασίσαμε ότι θα αναπέμψουμε το θέμα συζήτησαν οι συντονιστές και στο τέλος αυτής της ε, συζητήσεως διατηρήσαμε μέχρι την 31 Μαΐου την ημερομηνία για τροπολογίες όπως διαβεβαίωσα θα έχουμε τις μεταφράσεις ε, μέχρι το, ε, τη συνεδρίαση του Μαΐου τον ε, Μαΐο κατά τρόπον ώστε να έχουν όλοι τα αναγκαία στοιχεία και να μπορέσει και ο εισηγητής να προχωρήσει για να μην φτάσουμε στον Οκτώβριο του προωθηθεί το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τις ε, ανακοινώσεις ε, του Προέδρου έχω τον κύριο Κράμερ που ζήτησε τον λόγο. Ο κύριος ε, Κράμερ λέγει ότι εδώ υπάρχουν στα πρακτικά υπάρχει μια ημερομηνία άλλη από αυτή που συζητήσαμε χθε που ήταν 10 Μαΐου. Αντιλαμβάνουμε ότι όλες οι μεταφράσεις θα είναι έτοιμες μέχρι τις 10 Μαΐου. κάποιος άλλος, άλλο θέμα, είσαστε όλοι ευτυχείς ή κάπως τέλος πάντων ικανοποιημένοι με αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Και προχωράμε τώρα στις ψηφοφορίες. Has everybody got their voting machines? I know. Ε, ξέρω ότι έχετε όλοι τα μηχανήματά σας. Ο κύριος Μπέρκ ε, είναι νέος και γι' αυτό ε, κάθε φορά ο κύριος Μπέρκ θα μπορεί να ψηφίσει διαχειρός ενώ οι άλλοι θα πρέπει να ψηφίσουν με την κάρτα τους παρακαλώ κάντε μία δοκιμή για να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θα ψηφίσουν σωστά ξεκινά η δοκιμαστική ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Για δέστε ποιος, ποιος κέρδισε πέραν του κυρίου Μπέρκ. Ο κύριος Μπέρκ φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως θα ψηφίζει σύμφωνα με την δική σας ε, ε, ε, τις δικές σας οδηγίες. Ανήκει, έχετε κάποιον αντικαταστάτη ένα μέλος αναπληρωματικό εδώ. Παρακαλώ τότε αυτό το αναπληρωματικό μέλος να μην ψηφίζει. Γιατί είστε υπεράριθμοι. Ροβινιέτ. Είμαστε έτοιμοι. Τροπολογία 41. Ε, ξεκινάμε με την κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 αποσύρεται. 10 του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 με την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 και 46 μαζί, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο και για τις δύο μαζί. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Μπέρκε, ε, εσείς είσαστε υπέρ, μάλιστα. Λίγη η ψηφοφορία. 21 ε, υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 48, 49 και 50 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 ε, του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 51 καταπίπτει 52 αποσύρεται 53 και 54 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58, 59 και 60 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 12 ε, του εισηγητή υπέρ. Με συγχωρείτε, ε, καταπίπτει. Και πάμε τώρα στην 65. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 του, 13 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Η 67 καταργείται όπως και η 68 και πάμε τώρα στη 15 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 με την προφορική τροπολογία. Ε, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία και ο κύριος Μπέρκερ είναι υπέρ. 15 υπέρ, 22 κατά, απερίφθη. 73-74 ε, σε δύο τμήματα. Το πρώτο μέχρι το is to be used και το δεύτερο to reduce the negative impact of transport. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Ας κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά ας επαληθεύσουμε. Κλείνει. Ε, 18 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 75 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 και 77 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 αποσύρεται και τώρα ερχόμαστε στη 18 του εισηγητή με την προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83. Α, κατέπεσε. Όπως και η 80, η 81, 84 και πάω στην 85. Θα τα καταφέρω. Πού θα πάει ώσπου να φύγω. Ε, κατά. Αποχές. Ε, μόνο εάν πω ότι απερίφθη έχει απορριφθεί. 86 της κυρίας Τικάου. Καταπίπτει 19 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 και 89 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται 91 ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη 92 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 και 95 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 26 υπέρ, κατά, αποχές. Ας κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο για την 26, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. 19 υπέρ, 15 κατά, άρα εγκρίθηκε. 97 του κυρίου Λάιχτριντ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 99 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίθηκε 18 υπέρ, 17 κατά. Η 100 ε, της κυρίας Λίχτενμπέργκερ. Είναι διαφορετικό το θέμα, δεν καταπίπτει. 100 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ. Κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 100 της κυρίας Λίχτεμπέργκερ ξεκινά. Κύριε Μπέρκε. Λίγοι. 18 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. 101 της κυρίας Λίχτεμπεργκερ, Κατά αποχές απορρίπτεται 28 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 καταπίπτει 103 της κυρίας Λίχτενβέργκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 και 30 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 33 ε, Τη κυρίας Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δύο του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 πρέπει να ψηφίσουμε ακόμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 και 38 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 ε, 9 ε, ναι, υπέρ κατά αποχές και τώρα το σύνολο του, ε, της συστάσεως ο κύριος Μπέρκε είναι ε, υπέρ ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι λίγοι 27 υπέρ, 1 κατά, 11 αποχές. Συγχαίρουμε, συγχαίρουμε τον εισηγητή κύριο Αλκαντράουι. Okay, change of shift on the top table. Ωραία. Αλλάζουμε βάρκια εδώ πέρα, στο Προεδρείο. Περνάμε στην έκθεση Κουμουτσάκου για την ανάπτυξη μιας, ε, περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Πρώτη ψηφορία. ξεκινάμε. Άρθρο 1, συμβιβαστική λύση α Θα δούμε πρώτα τη συμβιβαστική λύση και μετά την προφορική τροπολογία. Α, πρώτα την, πρώτα την προφορική τροπολογία πρέπει να κάνουμε. Πρώτα η προφορική τροπολογία αντικαθιστούμε το economic growth με το economic resilience. Υπέρ. Κύριος Κομουτσάκος. Uh, Δεν είμαι υπέρ αυτή τη προφορική τροπολογία, σα το λέω πληροφοριακά. Ο εισηγητή είναι κατά τη προφορική τροπολογία. Αυτό είναι επίσημη αντίρρηση του ΕΛΚ. Θέλετε να ψηφίσουμε. Ωραία, ναι. Αν θέλετε να ψηφίσουμε, οκ. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία να αντικατασταθούν λέξεις economic growth από το economic resilience. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται η προφορική τροπολογία και περνάμε στο αρχικό κείμενο της συμβαστικής πρότασης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C. Τα άλλα καταπίπτουν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Ι, e. υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με τις υγιές σας. Συμβαστική τροπολογία G, υπέρ. Κατά, αποχή, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Και εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Ε, προτείνω... Φαντάζομαι ότι θα καταψηφιστεί, αλλά πρέπει να την ψηφίσουμε. Είναι η ίδια με πριν. Ψηφίζουμε την, την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, στη συμβαστική τροπολογία H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία I υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. MV3 στο άρθρο 2α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Νομίζω πρέπει να περάσουμε στην 53 τώρα. Τροπολογία 53 ως προστίκη. Υπέρ. Λέει, αν η συμβαστική τροπολογία C εγκριθεί, που εγκρίθηκε, προς, την ψηφίζουμε ως προστίκη. Υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τροπολογία 53, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Next is 56. 56 του κύριου Τέιλορ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 57 άρχεται η ψηφοφορία Everybody voted. Vote is closed. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 59 καταπίπτει 63 του κυρίου Τέιλορ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά MV6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 καταπίπτει, ό, έχει αποσυρθεί έτσι κι αλλιώς. Περνάμε στη Ρέτζι 15 επί του άρθρου 2 δέλτα α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 71 του κ. Τέιλορ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 Wills υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 του εισηγητή συμπίπτει με, το, ε, με την MV11 είναι ταυτόση με την MV11 στο άρθρο 3 συγκεκριμένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 Ρέτζι Ρέτζι 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε κατευθείαν στη Ρέτζι 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμβη 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 Τέιλορ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. «92» της κυρίας Βίλς στο 32α υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για 92 άρχεται η ψηφοφορία. is Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ΠΕΣ 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήταν η ΠΕΣ, ΦΙΣ, 22. 90, Βαντάλεν. Βαντάλεν, 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 90, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μετά 99 και της κυρίας Wills. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 του κ. Τέιλορ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 της κυρίας Βίλς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φύση 29 πες 29 υπέρ κατά αποχές 16 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Z, άρθρο 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πες 36 υπέρ κατά απορρίπτεται Μιλάνα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κύριος Βαντάλεν 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, προφορική ε, τροπολογία η οποία εγκρίνεται 113 Βίλς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πες 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 πες 41 και πες 42 και 44 ίδιες μαζί τις ε, εξετάζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 του κυρίου Τέιλορ. Ίδια με την ε, budget 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117. Με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στην έκτη της Επιτροπής Προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, budget 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 26 Ρέτζι το πρώτο κομμάτι χωρίς τις λέξεις Assess the Territorial Impact of the Program το πρώτο κομμάτι λοιπόν πρώτα της Ρέτζι 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα με τις λέξεις αυτές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το οποίο μας οδηγεί στην 27 ίδια με την 49, 51 και 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. και στην 28 τώρα, ίδια με την ΠΕΣ 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 μαζί με ΠΕΣ 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η υπαριθμόν 1 συμπίπτει με την ΠΕΣ 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική K, κάπα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 34 βίλς υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε λίγο την 34 της κυρίας Βίλς. Παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι λήξη ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 35 επίσης βίλης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 Τελευταία πρόταση που είναι προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 37 με την τελευταία πρόταση που είναι προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 3 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική L Είχαμε πρώτα την προφορική τροπολογία που ήταν η ίδια με του Economic Resilience υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η L ως έχει υπέρ κατά εγκρίνεται. Ε, της κυρίας Φώστερ η 40 απορρίπτεται, Taylor 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 6 και πες 5 που είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας 8 μαζί με την ε, προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 ε, βίλς υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επομένως, Ρέτζι 7 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Ρέτζι 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πες 9. Όχι, ζητώ συγγνώμη. 44. Βλάστο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πες εννέα τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Budget 1 σε δύο μέρη με τις λέξεις when the program is reviewed υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Υπαριθμόν 6 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εποχές. κρίνεται Πες του 10. Όχι. Πίπτη. Ε, Ρέτζι 10 υπέρ. Κατά. εποχές Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία λοιπόν. Η πρόταση έτσι όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουν ψηφίσει όλοι. Λήξη ψηφοφορίας. 37 υπέρ, κανείς κατά και δύο αποχές. Το νομοθετικό ψήφισμα άρχεται η ψηφοφορία. Όλοι ψήφισαν. Κλείνει η ψηφοφορία. 36 υπέρ, κανείς κατά δύο αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Okay. Thank you for that. Σας ευχαριστώ. Όσοι θέλουν να φύγουν μπορούν να φύγουν ήσυχα ήσυχα. Παρακαλώ. coffee, Κύριε Κουμουτσάκο, μετά την ψηφορία βλέπω ότι επιθυμείτε διαπραγματευτική εντολή για να ξεκινήσετε συζητήσεις με τους σκιώδης και τον εισηγητή της Επιτροπής Αλίας με το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν για, την πρώτη, για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί να δοθεί αυτή η διαπραγματική εντολή επί τη βάση της υιοθετημένης θέσης. Όχι, έτσι. Okay. Έχετε αυτή την διαπραγματική εντολή κύριε Κουμουτσάκο και πάντοτε θυμίζω στους ηγητές μας ε, αυτή η εντολή είναι η εντολή την οποία αποφάσισε η Επιτροπή και θα πρέπει να κινηθείτε με βάση αυτή την εντολή. Κύριε Κουμουτσάκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Ελπίζω ότι τα αποτέλεσματα θα είναι θετικά. Σας ευχαριστώ πολύ όλους ξανά. Okay, colleagues, the next Πολύ καλά. Μετά που πάμε, νεράκι. Πίνουμε νεράκι. Επόμενο θέμα. Ε, οδηγία χρόνου εργασίας, εφαρμογή της ε, κοινωνικής νομοθεσίας στις οδικές μεταφορές, ανταλλαγή απόψεων. Εγώ είμαι ο, ο εισηγητής ως πρόεδρος. Να θέσω στο πλαίσιο της αυτή την έκθεση και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Σίλβερ της Κομισιόν να πάρει το λόγο και μετά τον κύριο Πασκαρέλη και θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Η Κομισιόν πολύ, πολύ πρόσφατα δημοσίευσε ένα εγγραφό για την αναθεώρηση της Γενικής Οδηγίας Χρόνου Εργασίας 2003-88 όπως και μια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού 561 ε, για τους χρόνους οδήγησης και ξεκούρασης ε, και την ειδική οδηγία χρόνου εργασίας ε, για τις οδικές μεταφορές, οδηγίες, 2015. Το 2007 και 2008 η Επιτροπή Απασχόλησης ήταν ως κύρια Επιτροπή αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει η ίδια αλλά ορισμένες πτυχές οδικών μεταφορών παίζουν ρόλο σε αυτά τα έγγραφα οι συντονιστέ μας στην Επιτροπή Μεταφορών αποφάσισαν να καλέσουν αντιπροσώπους ε, από την Κομισιόν για μια ανταλλαγή απόψεων. Η Κομισιόν ιδιαίτερως ε, προσκλήθηκε να <clears throat> ρίξει φως στις διάφορες δυνατότητες μεγαλύτερης εναρμόνισης των κανόνων ε, χρόνου εργασίας για όλους τους μετακινούμενους εργαζόμενους σε οδικές μεταφορές που αυτοί οι κανόνες συζητώνται αυτή τη στιγμή στην ε, αναθεώρηση της ε, οδηγίας, το πλαίσιο της αναθεώρησης οδηγίας χρόνου εργασία. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη, του κανονισμού χρόνου οδήγησης ε, και ξεκούρασης ε, και την ειδική οδηγία για το χρόνο εργασία τη 15.002, η Κομισιό, ζητήθηκε από την Κομισιόν σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων να σχολιάσει τα εξή θέματα. Πρώτα, τις θετικές πτυχές όπως επίσης και τα προβλήματα στην τρέχουσα ε, εφαρμογή της του κανονισμού και της ε, οδηγίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεύτερον, πώς τα κράτη-μέλη ε, πληρούν τις υποχρεώσεις αναφοράς που έχουν και ποια κράτη-μέλη ακόμα πρέπει να βελτιώσουν την θέση τους σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτό το θέμα. Τρίτον, ποιοι είναι οι λόγοι για τις σημαντικές αποκλήσεις στη συχνότητα παραβάσεων ε, που συλλαμβάνονται στα διάφορα κράτη-μέλη, που εντοπίζουν τα κράτη-μέλη και τέταρτον τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στην εφαρμογή ε, του ψηφιακού ταχυγράφου. Όπως σας είπα έχουμε μαζί μας δύο εκπροσώπους της Κομισιόν, τον κύριο Σίλβερ από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και τον κύριο Πασκουαρέλη από τη Γενική Διεύθυνση MOVE. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα τους δώσω το λόγο για να ξεκινήσουν αυτή την ανταλλαγή απόψεων επί τη βάση των αρχικών μου παρατηρήσεων. Μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη. Κύριε Σίλβερ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών. Έχετε το λόγο. <clears throat> Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που στείλατε στην Κομισιόν να εξηγήσουμε το στάδιο των ασιών σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των κανόνων χρόνου εργασίας. Το θέμα είναι περίπλοκο. Ο χρόνος εργασίας για τους οδικούς μεταφορείς είναι περίπλοκο διότι διέπεται από τρία διαφορετικά νομικά κείμενα. Την Γενική Οδηγία Χρόνου Εργασίας ε, που περιλαμβάνει γενικούς κανόνες. Ε, ο κ θα, ε, θα, αυτή θα τη σχολιάσω εγώ και ο κ. Πασκορέλη τι πιο ειδικέ οδηγίες. Ε, η 2003-88 το 88 καθορίζει λοιπόν γενικούς κανόνες για μέγιστους ε, εβδομαδιαίους χρόνους εργασίας, ε, ημερήσιες και εβδομαδιαίες ε, ώρες ξεκούραση, άδειε κλπ. Όμως περιλαμβάνει και ένα μεγάλο αριθμό παρεκκλήσεων καθώς επίσης και προβλέψει ελαστικότητας. Το πεδίο εφαρμογής είναι πολύ πλατή, καλύπτει όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις εργασιακές δραστηριότητες, σε όλη την Ευρώπη εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ειδικές, ε, ειδικοί κανόνες χρονορασίας ε, δυνάμει άλλων νομοθετικών κειμένων. Αυτή είναι και η περίπτωση των οδικών μεταφορών και των αεροπορικών μεταφορών. Ε, ε, καλύπτονται από αυτή το τομή, καλύπτονται από ειδικέ οδηγίε, το ίδιο και με τι ε, νέες μεταφορέ, που ε, στηρίζονται σε, ε, είναι οδηγίε του Συμβουλίου κατόπιν διαπραγμάτευση στου κοινωνικού φορεί. έχουμε τον κανονισμό 561 του 2006 για τις οδικές μεταφορές με διαδικασίες εναρμόνισης, με, κανόνες εναρμόνισης ε, για τους χρόνους εργασίας και ξεκούρασης και την οδηγία 15.002 για το συνολικό χρόνο εργασίας που περιλαμβάνει και τους αυτοαπασχολούμενους. Ε, έχουμε τρεις κατηγορίες ε, οδικών μεταφορέων οι οποίες εξαιρούνται των διατάξεων του, των ειδικών αυτών κειμένων και καλύπτονται συνεπώ μόνο από τη Γενική Οδηγία Χρόνου Ρασία. Αυτοί είναι οι κινούμενοι εργαζόμενοι στα οχήματα μικρότερων των 3,5 τόνων, ε, εργαζόμενοι σε οχήματα ε, που ε, μεταφέρουν λιγότερους από 10 επιβάτες και εργαζόμενοι σε συνήθεις ε, ε, υπηρεσίες μεταφοράς που καλύπτουν αποστάσεις μικρότερες των 50 χιλιόμετρων. Τώρα, αυτή, αυτή η οδηγία αναθεωρείται, είναι υποαναθεώρηση αυτή τη στιγμή. Η προηγουμένη αναθεώρηση της οδηγίας ε, είχε λήξει με αποτυχία το 2009 και η Κομισιόν είχε από τότε ε, ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία αναθεώρησης οδηγίας. Οι στόχοι της αναθεώρησης είναι εξή. Πρώτον, να ε, προσαρμοστεί προσαρμοστούν αυτοί οι κανόνε σε, ε, σε μια νέα πραγματικότητα και στις απόψει των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων να μειωθεί η νομική ασάφεια και να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα που προέκυψαν από την ομολογία του ε, δικαστηρίου. Ε, επίσης έχουμε ορισμένα προβλήματα εφαρμογής σε κάτι μέλη τα οποία θα πρέπει επίση να ρυθμίσουμε. Ξεκινήσαμε την διαβούλευση τον περασμένο Μάρτιο με μια πρώτη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ζητήσαμε τους κοινωνικούς εταίρους, τους, τους, εταίρους να μας ε, πούν τη γνώμη τους σε ό,τι αφορά την ανάγκη και το εύρος μιας α, προσαρμογής. Ε, μετά το Δεκέμβριο του περασμένου τους ξεκινήσαμε μια δεύτερη, το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης και ταυτόχρονα δημοσιεύσαμε και μια έκθεση εφαρμογής ε, όπου εντοπίζουμε τα νομικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί με την εφαρμογή της ε, οδηγίας μέχρι τώρα ταυτόχρονα δημοσίευσαμε και μια οικονομική και κοινωνική μελέτη ενός εξωτερικού συνεργάτη συμβούλου που εντοπίζει τα βασικά οικονομικά και κοινωνικές, βασικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της οδηγίας. Θέλαμε να δώσουμε λοιπόν στους κοινωνικούς εταίρους όλα τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, στις απαντήσεις τους. Πήραμε απαντήσεις, πάνω από 40 συγκεκριμένα απαντήσεις μέχρι την περασμένη εβδομάδα τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι απαντήσει των κοινωνικών εταίρων. Τα βασικά συμπεράσματα τα οποία μπορούμε ήδη να βγάλουμε από τη δεύτερη διαβούλευση είναι τα εξή. Πρώτον, οι κοινωνικοί εταίροι καλωσορίζουν τη δημοσίευση των αναλυτικών εκθέσεων, θεωρούν το ανακοίνωση της Κομισιόν χρήσιμη, λένε ότι εντοπίζουν τα βασικά, εντοπίζει τα βασικά σημεία αναθεώρησης, ε, ε θεωρούν ότι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για να βρουν καταλήγουν σε συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα σχετικά με το χρόνο εργασία που έχουν παρουσιαστεί από την, ε, όλο αυτόν τον τελευταίο καιρό και ε, οι βασικοί κοινωνικοί εταίροι διατομιακοί έχουν εκφράσει την προθυμία τους να διαπραγματευτούν μεταξύ τους για να βρουν κοινές, κοινώς αποδεκτές λύσεις. Βέβαια πρέπει να γνωρίσουμε ότι το σημείο αφετηρίας ε, διαφέρει από κοινωνικό εταίρο σε κοινωνικό εταίρο, τόσο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των ε, διαπραγματεύσεων, το πεδίο εφαρμογή δηλαδή, όσο και ε, τις βασικές τους θέσεις σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Ε, υπάρχουν όμως ε, συνθήκες για έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων που θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια κοινή δήλωση βέβαια όλων των κοινωνικών εταίρων ότι επιθυμούν να ξεκινήσει η διαπραγματεύση αυτή. Συνεπώ, βρισκόμαστε στην περίοδο κατά τη διάρκεια τη οποία η Κομισιόν θα πρέπει κατά βάση να περιμένει απόφαση από πλευρά των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημε διαπραγματεύσει. Τώρα, ποια είναι τα βασικά ζητήματα υπό διαπραγμάτευση, ε, στην, αυτά δηλαδή τα οποία θέσαμε στη δεύτερη ε, διαβούλευση. Εμεί είχαμε πει ή να εστιαστούμε στα ζητήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί δυσκολίε στην εφαρμογή της ισχύουσας νομολογίας ε, παράδειγμα το πώς μετράται ο χρόνος εργασίας, ε, το πώς υπολογίζεται σε ε, περιπτώσεις ε, βάρδιας σε δημόσια νοσοκομεία κλπ. Και τις, το χρόνο ξεκούρασης που δίδεται σε περιπτώσεις υπέρβαση του χρόνου εργασίας. Αυτή ήταν η μία αναλυτική λύση που προτείναμε. Η δεύτερη αναλυτική λύση που, είπαμε, που προτείναμε ήταν μια ανακληση που προτειναμε η δευτερη ανακληση που ειπαμε που προτειναμε προσθέτοντας και άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα διατάξεις για την βελτίωση καλύτερης ισορροπίας εργασίας προσωπικής ζωής, ε, η ρήτρα αυτοεξαίρεσης, το θέμα των αυτοπασχολούμενων εργαζόμενων, τι γίνεται με τους εργαζόμενους που έχουν πολλές θέσεις εργασίας παράλληλα, πώς θα πρέπει να προσμετάλλεται σε αυτούς ο χρόνος εργασίας και ευελιξία, ε, πρόσθετη ευελιξία. Ιδιαίτερα για τις οδικές μεταφορές αναγνωρίζουμε ένα θέμα το οποίο είναι σίγουρα ανοιχτό. Όπως σας είπα έχουμε κάποιες κατηγορίες ε, μετακινούμενων εργαζόμενων στις οδικές μεταφορές που δεν καλύπτονται από, τις, ε, από τα ειδικά νομοθετικά κείμενα καλύπτονται από τη γενική οδηγία. Όμως, αυτή η γενική οδηγία εφαρμόζεται σε αυτούς, Εφαρμόζεται σε αυτούς, αλλά όχι οι ποσοτικοί κανόνες που εφαρμόζονται σε άλλους κανόνες, σε άλλους εργαζόμενους σε ό,τι αφορά ε, χρόνο ξεκούρασης και τη νυχτερινή εργασία. Η γενική οδηγία έχει κάποιες διατάξεις οι οποίες χρήζουν ερμηνείας κάθε φορά και ε, ε τους ερμηνεύουν τα κράτη-μέλη με πολύ διασταλτικό τρόπο υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, δεν χορηγείται επαρκής βαθμός προστασίας σε αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι καλύπτονται μόνο από τη γενική οδηγία. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το χρόνο ξεκούραση και τη νυχτερινή εργασία. Συνεπώ, υπάρχει θέμα με αυτού. Ε, αν θα πρέπει δηλαδή να εναρμονιστούν οι όροι για αυτού του εργαζόμενου ε, σύμφωνα με τα όσα ε, ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους ε, δυνάμει της οδηγίας 2002 του 2015. ε, ε, περιμένουμε από τους ε, ε, κοινωνικούς εταίρους να μας πούν τη γνώμη τους. Τα συνδικάτα τίνουν να είναι υπέρ της συνολικής εναρμόνισης, αλλά οι απαντήσεις ήταν ε, πολύ ολιγόλογες, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουν μεταξύ του οι κοινωνικοί εταίροι, αν θα αποφασίσουν συνολική προσαρμογή ή σε συγκεκριμένα λίγα ζητήματα. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Πασκορέλη θέλει να προσθέσει κάτι. Ε, δεν είναι τόσο να προσθέσω, Πρόεδρε. Όσο να απαντήσω τα τέσσερα ερωτήματα που πιο συγκεκριμένα ετέθησαν για τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και κινητικότητας που είναι υπεύθυνη για ένα άλλο σετ κανόνων για τον κανονισμό 561 για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης η οδηγία εφαρμογής που συνοδεύει τον κανονισμό και μετά η συγκεκριμένη οδηγία για τους μετακινούμενους εργαζόμενους όπως είναι οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων. Εμείς πιστεύουμε και θα, έχω τις, θα λάβω τις, και τις ερωτήσεις σας για τα υπέρ και τα κατά του πακέτου αυτού του νομοθετικού ότι η κοινωνική νομοθεσία είναι θεμελιώδες εργαλείο για να προφυλάξουμε τρεις στόχους. Ασφάλεια, οδική, δίκαιο ανταγωνισμό και κατάλληλες συνδικές εργασίας σε κάθε τομέα. Οι κανόνες αυτοί ε, για το χρόνο οδήγηση ισχύουν από το 1985. Ο 561 του 6 ε, εξυγχρόνησε την νομοθεσία που υφίσταται από το 85 και συνοδεύτηκε από μια οδηγία εφαρμογής την 22 του 2006 με την, ε, με την οποία εισάγαμε τον ηλεκτρονικό ταχυγράφο που είναι πολύ πιο ακριβής από τον αναλογικό ταχυγράφο, τον ψηφιακό. Και είχαμε και την ε, έγκριση της οδηγίας 15 του 2000. Τώρα, όλα αυτά εξαρτώνται από την συμμόρφωση με τους κανόνες και από μια αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των θετικών τυχών, των υπέρ, πέραν το ότι δηλαδή υφίστανται οι κανόνες και είναι κοινοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απλοί και εύχριστοι... οι παλαιοί κανόνες δηλαδή του 85 και έχουν και μια απαραίτητη ευελιξία μέχρι ένα βαθμό. Ο νομοθέτης λοιπόν προεκτείνει την ευθύνη συμμόρφωση με τους κανόνες όχι μόνο στον οδηγό, αλλά και σε όλη την αλυσίδα τη διοικητική. Τον μεταφορέα, τον εκφορτωτή κτλ. Και συνεργάζεται με τις εταιρείε κατά τρόπον ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες και να υπάρχει ευθύνη, να υπάρχουν και κυρώσεις για τις οποιασδήποτε δηλαδή, ε, για τα οποιαδήποτε παραπτώματα. Η Κομισιόν προάγει μια εναρμονισμένη ερμηνεία και η εφαρμογή των κανόνων αυτών σε όλο το έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κάνουμε από κοινού με μια επιτροπή από εκπροσώπηση των κρατών μελών, επιτροπολογία, έχουμε την Επιτροπή Κοινωνικών Κανόνων, που αποτελείται και πάλι από εκπροσώπους των κρατών μελών, όπως έλεγα, όπου παρίστανται και κοινωνικοί εταίροι και ενδιαφέρομενα μέρη. Ε, οι εκπρόσωποι των ε, συνδικάτων, και εκπρόσωποι των ε, ρυθμιστικών αρχών και των αρχών εφαρμογής στα διάφορα κράτη-μέλη και προχωρούμε με το εφαρμοστικό έργο του κανονισμού που δεν είναι μόνο η οθέτηση εφαρμοστικών κανόνων από καιρού καιρών αλλά και κοινή ερμηνεία και κοινέ συστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε έξι σημειώματα καθοδήγηση αν θέλετε που δεν είναι δεσμευτικά αλλά δίνουν την ερμηνεία η οποία προσφέρεται από την Κομισιόν προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κάποια από τα πιο δύσκολα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της, ε, του κανονισμού χρόνου Έχουμε συγχρηματοδοτήσει και το πρόγραμμα TRACE, πρόγραμμα επιμόρφωσης ε, σε συνεργασία με, όλους, με όλα τα υπεύθυνα γραφεία εφαρμογής. Ένα άλλο πρόγραμμα ε, συνεργασίας των αστυνομικών αρχών που αποσκοπεί στους κοινού ε, κανόνες ε, προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους, για τους αξιωματικούς και μετά έχουμε πρωτοβολία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, την, για τον κανονισμό 561 όπου έχουμε εξαγάγει τα δικά μας πρότυπα χρόνου εργασίας στην ευρύτερη ευρασιατική περιοχή μέσω του, της συμφωνίας AETR υπό την αιγίδα της ε, συνεργασίας ε, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων για να έχουμε από τον Ατλαντικό στο Βλαδιβοστόκ ενιαίους κανόνες αν θέλετε. Εκρεμούν ακόμα κάποια θέματα που θα πρέπει να καλυφθούν για να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια σε όλη τη διοικητική αλυσίδα ώστε να οργανώνονται οι επιχειρήσεις κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των οδηγών. Έχουμε διαφορετικές δυνατότητες. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποίησεις μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Και υπάρχουν και κάποιοι, και κάποιοι έλεγχοι που είναι αρκετά αποσπασματικοί το πεδίο αντί για συστηματικούς ελέγχους στα κέντρα, στις ε, έδρες των επιχειρήσεων γιατί έχουν αργήσει οι επιχειρήσεις ε, να συστήσουν ένα σύστημα ε, αξιολόγησης του κινδύνου ώστε να βαθμολογούνται οι επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην συμμορφώνονται με τους κανόνες. ώστε να πρημοδοτούνται, αν θέλετε, αυτοί που συμμορφώνονται. Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή αυτή, από την έκθεση της κυρίας Ράνερ ε, του 2009, ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα διάφορα κράτη-μέλη για την ίδια κατηγορία παρατομάτων ε, ε, αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους. Και αυτό είναι, ένα, είναι αντικειμενικά ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και σε σχέση με το οποίο δεν είχαμε μέχρι τη στιγμή τα μέσα διάθεσή μας και είχαμε και αποκλίνουσε αρμοδιότητες μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ε, επιβολή του νόμου και τις όποιες ποινικέ κυρώσεις που θα μπορούσαν επίσης να υπάρχουν σε μερικές περιπτώσεις. Είχαμε διαμαρτυρίες λοιπόν για έλλειψη εναρμόνισης ε, των κυρώσεων η οποία προκαλούσε στρέβλωση του αναγωνισμού και θα ήθελα να είμαι σαφίστατος επ' αυτού. Δεν πρόκειται για την διαφορετική εφαρμογή των κυρώσεων. Πρόκειται για την μη συμμόρφωση προς τους ε, κανόνες που προκαλεί στρεβλώσεις. Δεν είναι θέμα ισότιμης μεταχείρισης. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι θέμα ίσης και ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου και ίση εφαρμογή των κυρώσεων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικό πρόβλημα διότι η Ένωση στο σύνολό της μέχρι στιγμή, δεν είχε τα μέσα στη θέση τη και την αρμοδιότητα για να το κάνει. Τώρα ελπίζουμε θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέσω της ε, ευρύτερης, ε, του ευρύτερου φάσματος αρμοδιοτήτων που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Για την 15 τώρα ε, οδηγία για τους ε, εργαζομένους, τους μετακινούμενους, ο συνάδελφος ε, Σίλβα είχε παρουσιάσει τα γενικά στοιχεία λίγο νωρίτερα, αλλά εδώ έχουμε, αν θέλετε, ένα κοινωνικό νομοθέτημα. Αφήνω στην άκρη τα λεπτά ζητήματα πεδίου την εφαρμογή τους αυτοαποσχολούμενου, για παράδειγμα που συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία αυτή και όχι στη Γενική Οδηγία Χρόνου εργασία, η διαφορά των δύο νομοθετημάτων είναι μικρή και κυρίως όπως είπε ο κύριος Σίλβα μιλούμε κυρίω για τις διατάξεις της νυχτερινής εργασίας που ε, δεν υφίστανται στην ε, Οδηγία Μεταφορών αλλά εδώ καλύπτουμε το 70% ε, του αυτοαποσχολούμενου ή μισθωτού εργαζόμενου οδηγού και το οποίο σε σχέση με την ε, DG Move ε, εξαρτάται από, την, από τη σύγκρισή της με τους γενικότερους κανόνες μετακινούμενης εργασίας και οδήγησης. Έχουμε μια, κάποιες διαδικασίες παρακολούθησης και έχουμε το θέμα του, το βασικό θέμα ότι ο νομοθέτης εφαρμόζοντας την οδηγία 2062 μαζί με την οδηγία χρόνου οδήγησης 2006 αποφάσισαν να μην προεκτείνουν την ε, εφαρμογή επιβολής ώστε να καλυφθεί και η οδηγία του 2002 γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με την σωστή εφαρμογή τα κράτη-μέλη, αλλά η παρακολούθηση και η επιτήρηση είναι δυνατή μέσω διοικητικών ελέγχων και των ταχυγράφων. Κάποιοι όμως αυτό οι οδηγοί δεν έχουν το ενδιαφέρον να καταχωρήσουν όλες τις δραστηριότητες τους ως λυπή εργασία. Μόνο η οδήγηση μπορεί να καταγραφεί από τους ταχυγράφους, ενώ όλες οι λοιπές δραστηριότητες εξαρτώνται από την ε, καλή θέληση, αν θέλετε, την καλή πίστη των ε, οδηγών. Εμένως υπάρχει αυτό το θέμα των καταγραφών. Είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Πρόεδρος, αλλά έχουμε μακρύ κατάλογο μιλητών και προσπαθώ να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία θέσατε κύριε Πρόεδρε. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχουμε μία μακριά συνεδρίαση, έχουμε καθυστερήσει ήδη και μπορώ να ελέγξω πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά όχι όλα και γι' αυτό προσπαθώ να σας καθοδηγήσω. Δηλαδή αντιλαμβάνουμε ότι χρειάζεται πιο σύντομες απαντήσεις. Μου είπατε αν έχουμε καλύψει τις ε, υποχρεώσεις ε, για την υποβολή στοιχείων. Δεν πάμε πολύ καλά είναι η απάντηση. Τα κράτη-μέλη καθυστερούν να υποβάλουν τις απαντήσεις. Στο τέλος έχουμε ορισμένες διαδικασίες παραβίασης και για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τη συνολική μας έκθεση χρειαζόμαστε τις ε, απαντήσεις των κρατών ομοιογενώς, πράγμα το οποίο δεν διαθέτουμε πάντοτε. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, γιατί ε, εάν τα κράτη-μέλη δεν μας απαντούν και διότι ε, αυτή η οδηγία δεν είναι τόσο ομαλή όσο η οδηγία για το χρόνο οδήγησης όσον αφορά τις παραβιάσεις μεταξύ κρατών μελών. Υπάρχουν. Ε, υπάρχει μια συχνότητα στην οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που με τη σειρά τους εξαρτώνται από την διοικητική δυνατότητα η οποία αλλάζει πολύ από το ένα κράτος στο άλλο και από την ε, ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου ή όχι. Γιατί όπως σας είπα ότι αν υπάρχει ένα σύστημα βαθμολόγησης του κινδύνου επιτρέπει στα κράτη να επικεντρωθούν στα θέματα όπου είναι πολύ πιθανότερο να υπάρξουν παραβιάσεις από ό,τι αλλού. Τέλος, όπως σας είπα υπάρχει ε, ένα ε, πρόγραμμα ηλεκτρονικό το οποίο είναι έξυπνο και μπορεί να ενημερώνεται ε, με τις αλλαγές που υιοθετεί μέσω Επιτροπολογίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε τώρα έχουμε δύο μορφές του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να δούμε πόσο, κατά πόσο είναι αξιόπιστος να δούμε τα υπέρ και τα κατά και για να γίνει κάτι τέτοιο ετοιμάζουμε κάποια νομοθεσία η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια καταρτήσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται ουσιαστικά για μία εξέταση του παλιού κανονισμού του 1985 που θα παρουσιαστεί σαν ε, ε, νέος κανονισμός για το γονταχογράφο και θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο ελπίζουμε πριν το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Έχω εννέα ομιλητές στο κατάλογό μου και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ουσιαστικά θέματα που θέλετε να θίξετε αλλά θα παρακαλούσα να μην υπάρχουν επαναλήψεις ε, διότι όλοι δεν ακολουθούν τις ίδιες μεθόδους οπότε βοηθήστε με να επανακτήσουμε το χαμένο χρόνο. Ο κύριος Γκρός έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί στο Κοινοβούλιο για τις οδικές μεταφορές εδώ και χρόνια και όπου το θέμα της ρυθμίσεως στο παρελθόν ε, έχει προχωρήσει πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Επίσης υπάρχει μία πλειοψηφία επιχειρήσεων που συμφωνούν με τις απόψεις αυτές. Δηλαδή εάν εξετάσουμε τα προβλήματα δεν βλέπουμε ότι ο κάθε οδηγός φορτηγού είναι ένας δυνητικός εγκληματίας και δολοφόνος. Πρέπει να εξετάσουμε τα προβλήματα αλλά να τα εξετάσουμε εστιασμένα. Και αισθάνομαι ότι είναι θέματα τα οποία έχουμε ξαναδεί εδώ. Ε, διότι σε ορισμένες χώρες όπως ε, και στη δικιά μου χώρα δεν υπάρχει μία ουσιαστική πρόοδος ε, πρέπει να δούμε εάν οι έλεγχοι γίνονται στο δρόμο ή στην επιχείρηση έχουμε κάνει προτάσεις και βλέπουμε πώς προχωρούν ορισμένα κράτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προτάσεις για ορισμένα θέματα θέματα και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις εντός της χώρας οι οποίες μορφώνται και άλλες όχι. Τέλος, όσον αφορά την εναρμόνιση ε, των εθνικών οδικών μεταφορών και των υπερεθνικών, ε, εγώ δεν συμφωνώ ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα μπορούσαν, εφόσον αντιδρούν στις προτάσεις τις οποίες διατυπώνουμε. Δεν θέλουμε μεν όλα να είναι τέλεια αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια εναρμόνιση των ποινών σε σοβαρές περιπτώσεις ε, όσον αφορά τους ε, ελέγχους τους έχουμε επίσης επισημάνει δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε σε έναν ε, φορτηγατζή ότι δεν σέβεται τον χρόνο εργασίας εάν δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει από συγκεκριμένα θέματα τα, από συγκεκριμένε περιοχές σε ορισμένες ώρες. Βέβαια υπάρχει και το θέμα του ταχογράφου ο οποίος δεν λειτουργεί και στην περίπτωση αυτή ε, μπορεί κανείς ε, να το να δρανοποιήσει. Το ξέρουμε και εμείς, το ξέρουν και οι επιχειρήσεις. Οπότε θα παρακαλούσα αφενός να υπάρξει μία εφαρμογή πιο ενιαία στο εθνικό επίπεδο. Τρίτον, ε, δεύτερον να εξετάσουμε κράτος κατά κράτος και τρίτον αυτό που μας απασχολεί είναι οι διεθνείς μεταφορές. Δεν είναι δυνατόν σιγά σιγά οι παραδοσιακές επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται τα, τις αποφάσεις οι οποίες ε, πρέπει να ε, ανταγωνιστούν ε, επιχειρήσεις τρίτων χωρών οι οποίες κάνουν θέμητο ανταγωνισμό και καμποτάζ και παραμένουν στην Ευρώπη για δύο-τρεις μήνες και μετά γυρίζουν στη χώρα τους με ένα πάρα πολύ χαμηλό μισθό πολύ χαμηλότερο από ό,τι πληρώνουμε στην Ευρώπη. Πρέπει, δεν χρειάζεται εκεί να κάνουμε μελέτες, ε, να βρούμε λεπτομέρειες, αλλά να κάνουμε αμέσως ε, κάποια συζήτηση για την εφαρμογή των διατάξεων κατά τρόπον ώστε να αρθούν τα προβλήματα αυτό. Διαφορετικά θα χρειαστεί να ξεχάσουμε και να εγκαταλείψουμε τις εθνικές επιχειρήσεις ε, που είναι παραδοσιακές και δουλεύουν σωστά σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον, ε, ε, ε, την Επιτροπή για την Εισαγωγή και είναι βασικό να μπορέσουν να εξαφανιστούν οι κακοί μαθητές από το σύστημα για να μπορούν όλοι να λειτουργήσουν σωστά. Θεωρώ λοιπόν ότι η εφαρμογή του κανονισμού 561 να ε, επιτρέπει να υπάρχει μια πιο ενιαία εφαρμογή στις διάφορες χώρες αλλά εδώ πρέπει να επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει και να ζητήσει από τις χώρες που δεν εφαρμόζουν το σύστημα να απολογηθούν διότι το σύστημα διαφέρει πάρα πολύ Ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον καμία διασύνδεση με το οικονομικό σύστημα της ε, χώρας και πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να διοχετεύσουμε όλα αυτά σε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι μέτρα θα πάρετε. Αναφερθήκατε σε μία Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων που θα είναι πολύ χρήσιμη γιατί υπάρχουν ελάχιστες επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονται τις ε, συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να τις ελέγξουμε πιο συγκεκριμένα κατά τρόπον ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Αναφερθήκατε ε, και εις ε, τους ε, εργαζόμενους οι οποίοι διακινούνται σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας του χρόνου εργασίας και να αναρωτιέμαι εάν πρόκειται να, εφαρμογή, να ελέγξετε την εφαρμογή εντός των κρατών μελών διότι ξέρετε ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή παντού. Και διάβασα ότι θα υπάρξει ένας κοινωνικός κώδικας για τις μεταφορές, για τον κοινωνικό διάλογο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πότε μπορούμε να αναμείνουμε μια τέτοια πρόταση και τι θα περιλάβει. Αυτά είχα να πω σαν αφορά τις πρώτες ερωτήσεις μου και ζητώ συγγνώμη αλλά θα χρειαστεί να σας εγκαταλείψω άμεσα για αλλά ο συνάδελφός μου θα σημειώσει τις απαντήσεις. Αυτό πρώτο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα του χρόνου οδηγήσεως ε, για αποστάσεις κάτω των 50 χιλιόμετρων. Ξέρουμε ότι χρειάστηκε να αυξήσουμε αυτή την απόσταση στα 150 χιλιόμετρα για μικρές επιχειρήσεις, για αυτούς οι οποίοι οδηγούν μικρά φορτηγά και ε, ενδέχεται ε, ε, ένας μπογιατζής να μεταβεί σε 60-70 χιλιόμετρα για να κάνει κάποια δουλειά οπότε ήδη προ τριών ετών είχαμε εξετάσει το θέμα αυτό και διαπιστώσαμε ότι τώρα υπάρχει εξέταση του συγκεκριμένου σημείου διότι δεν θέλουμε να δυσκολεύουμε δυσκολέψουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη αλλά να τους διευκολύνουμε στην άσκηση των επαγγελμάτων τους. Επίσης ε, δύο φορές απέτυχε η συζήτηση ε, και στο θέμα του χρόνου ε, οδηγίας οδηγήσεως. Τους ελέγχουμε μέσω του τραχογράφου. Αλλά βέβαια το τι κάνει κανείς στην ιδιωτική του ζωή ε, στα πλαίσια των προσωπικών του μετακινήσεων είναι κάτι το οποίο ε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ε, ακόμη και αν ορισμένοι προσπαθούν να προβούν σε αλλαγές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είπαμε ότι αν υπάρχουν στρεβλώσεις του διαγωνισμού και τις διαπιστώσουμε και μπορούμε να τις εντοπίσουμε πρέπει να κοιτάξουμε να τις καταργήσουμε. Αναφέρομαι εδώ γενικά, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουμε και θα ήμουν ευτυχής αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να μας διατυπώσει προτάσεις. Επίσης στο τελευταίο σημείο μας είπατε ότι η εφαρμογή δεν είναι σωστή. Όλες οι χώρες συνένεσαν στο Συμβούλιο και βλέπουμε ότι εδώ όντως η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή έχει δίκιο να επικεντρώσει την προσοχή της όπου υπάρχουν πολλές παραβιάσεις και ε, να μπορεί κανείς να εφαρμόζει πιο απλές διατάξεις που διευκολύνουν και τον έλεγχο. Κύριος Κράμερ, και εγώ ευχαριστώ για την έκθεση, αλλά εδώ μιλάμε για την ασφάλεια στο δικό σύστημα και δεν πρέπει να διαχωρίζουμε μεταξύ των ε, ε, ελευθέρων επαγγελματιών και των υπαλλήλων και ε, θα ήθελα να θεωρήσω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τι κάνει κανείς αλλά ποιες είναι οι επιπτώσεις των πράξεων του. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα πιστεύω ότι αυτό δεν σρευλώνει τον ανταγωνισμό διότι ε, αυτό το στοιχείο περιλαμβάνεται σε όλα τα οχήματα τώρα αλλά δεν χρειάζεται αλλαγή. Όσον αφορά τους ελέγχους, ευχαριστώ το Ματιό που είπε ότι στη χώρα του υπάρχει το 2% το οποίο ζητήσαμε αλλά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι θευματοφύλακα των συνθήκων και πρέπει να παρακολουθεί τι κάνει εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να έχω κάθε χρόνο μία στατιστική και να υπάρχουν οι αυστηρότερες παραβιάσεις. Να ξέρω εάν υπάρχει μία αλλαγή από τη μια χρονιά στην άλλη στη συμπεριφορά κάποιας χώρας. Ε, εφόσον έχετε την κάλυψη του Κοινοβουλίου πρέπει να ενεργοποιηθείτε και ε, να μην ε, μας λέτε απλώς ότι τι έχετε κάνει εσείς αλλά και πώς απαντάτε στις δικές μας απαιτήσεις. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την road safety και ένα βασικό θέμα είναι η κόποση. Η ε, ε, κόποση, ναρκωτικά, ε, κατανάλωση ινοπνεύματος και η, είναι η κόπωση είναι ένα βασικό θέμα το οποίο πρέπει να ελέγχετε διότι διαφορετικά με τους ωραιότερους νόμους δεν θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε αύξηση της ασφαλείας. Επίσης έχουμε ελάχιστα σημεία στάθμευσης αλλά μειώνουμε ε, τους χρόνους γιατί αν υπάρχει ένα gigaliner, ένα τεράστιο όχημα θα χρειαστεί δύο θέσεις αντί για μία και εάν αυξήσουμε τις θέσεις σταθμεύσεως δεν πρέπει να είναι για τα τεράστια οχήματα αλλά για τα κανονικά. Μετά, όσον αφορά τη βλάβη του ταχογράφου, ξέρω ότι και ε, ε, ε, ταξιτζίδες ε, ε, μαστορεύουν τους ταχογράφους τους. Οπότε θα έπρεπε να εξετάσουμε αν υπάρχει παρεμβολή εγκληματική στο κλείσιμο ενός ταχογράφου. Ε, κάτι που θα σας εγγυωμένω δεν θα επαναλάβω πράγματα που έχουν ήδη λεχθεί. όταν, συζητάμε αυτό το, όταν συζητούσαμε αυτό το θέμα πριν από αρκετά χρόνια, ε, ήμουν, διαφωνούσα πλήρως ε, και κάθετα με την, Ευρω... με την υπάρξη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε αυτόν τον κλάδο και εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η γραφειοκρατία την οποία προκαλεί αυτή η νομοθεσία είναι τεράστια Εσεί γνωρίζετε, είστε Βρετανό, κύριε Πρόεδρε, ε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά τα νομοθετικά κείμενα έχουν δημιουργήσει ε, αρνητική διαφήμιση για την, Ευρωπα... στη... για την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ενωμένου από τότε που είχαμε την υπόθεση των ίσιων, ε, της ίσιας μπανάνας. και Ακούω μακροσκελείς παρουσιάσεις από τους εκπροσώπους Κομισιόν, τους άκουσα και αναρωτιέμαι σε ποιο πλανήτη ζουν. Διότι Σίγουρα είναι προφανές ότι δεν έχουν πρακτική γνώση του πώς εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες και τα προβλήματα που προκαλεί η εφαρμογή τους κυρίως στις ε, μικρές, ε, μικρές ε, και μεσές επιχειρήσεις, στους αυτοπασχολούμενους κλπ. Όταν είχαν προταθεί αυτά τα κείμενα και ιδιαίτερα το, το, το, το κοινωνικών κανόνων, είχαμε κάνει μια μελέτη ε, στην Ηνωμένο Βασίλειο με το κέντρο των επιχειρήσεων logistics και είχαμε 300 ε, τέτοιες επιχειρήσεις και μόνο στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Έκανα λοιπόν μια έρευνα και τους είπα και μάλλον ε, η οι που πήρα ήταν ακριβώς προ αυτή την κατεύθυνση ότι αυτά τα νομοθετικά κείμενα προσθέτουν γραφειοκρατία ήδη σε, σε ένα τομέα που ήδη χαρακτηρίζεται πολύ γραφειοκρατία και διοικητικά άκτη. Ε, και τώρα ακούω ότι γίνονται εκκλήσεις για ακόμα πιο αυστηρή νομοθεσία. Αυτά είναι πραγματικά παράλογα πράγματα. Ο εκπρόσωπος ε, της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης ε, μας έκανε κάποιες προτάσεις ότι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Να σας πω εγώ τι πρέπει να γίνει. Να μείνουμε και και να, να σας πω τι πρέπει να γίνει. Απλοποίηση και ελαστικότητα. Απλοποιήστε το διοικητικό άχθος, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοπασχολούμενους και ε, υιοθετήστε ευελιξία σε ό,τι αφορά το τι χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Διότι αυτό που προβλέπω εγώ είναι ότι αν διευρύνουμε και κάνουμε πιο αυστηρή την νομοθεσία θα βρούμε λύσεις σε προβλήματα που δεν υπάρχουν. Αυτό θα συστήνα εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας ξεκινήσουμε να εξετάζουμε πώς εμποδίζονται οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν, πώς εμποδίζονται οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που όλοι θέλουμε να κάνουν. Δηλαδή να μπορούν να δουλέψουν, να δουλέψουν όταν θέλουν και να ε, έχουν ένα λογικό εισόδημα στις μικρομεσαίες τους επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Μπακ. Ale They were. We try. Yeah, also The German Για τρίτη φορά μπορείς να ξαναξεκινήσεις, George. Όσον αφορά τους ελέγχους επιχειρήσεις θα ήθελα να σας πω ότι παλιά φωνάζαμε αλλά τίποτα δεν γινόταν. Αλλά στην έκθεση δεν αναφέρονται οι συνθήκες εργασίες που αναφέρονται στο οδικό απλό σύστημα. Δηλαδή ε, γιατί δεν καλύπτουμε όλους τους εργαζόμενους στις μεταφορές διότι λέγεται, ε, αναφέρεται αυτή η διασυνοριακή συμφωνία για τους σιδηροδρόμους η οποία έλυσε το πρόβλημα της ε, στρεβλωμένης σχέσεως αλλά δεν εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές και ουσιαστικά όσον αφορά τον ανταγωνισμό οι σιδηρόδρομοι ε, συναγωνίζονται τις οδικές μεταφορές και άρα θα πρέπει να ελέγξουμε το σύνολο. Αυτό όσον αφορά τους ελέγχους. Ε, κατά τη γνώμη μου τα ε, οχήματα κάτω από 3,5 νους θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπέψη και οι οδηγοί τους και ε, πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε συνήθως τους μικρούς επαγγελματίες αλλά θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τα χιλιόμετρα στα 50-60 από τα 15. Επίσης η υποχρέωση αναφοράς που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ένας εργαζόμενος ε, είναι πολυθεσίτης διότι αυτό πρόκειται, ε, αυτό είναι μία προσωπική συμφωνία μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη. Αν υπάρχουν σωστοί εποπτικοί μηχανισμοί τότε ε, θα να διαπιστώσουμε ότι πάντοτε θα υπάρχει μαύρη εργασία η οποία δεν ελέγχεται καθόλου, ιδίως σε ορισμένα κράτη και έχω πολλές επιφυλάξεις ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ε, ε, παράνομη μαύρη εργασία. Ευχαριστώ. Έχω τρεις ομιλητές ακόμη και θα πρέπει να είναι σύντομοι διότι προς το παρόν έχουμε καθυστερήσει 15 λεπτά η κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον κανόνα των, των αποστάσεων κάτω από 50 χιλιόμετρα. Τα κάποιος συνδικαλιστικά σωματεία επανειλημμένως μου έχουν πει ότι γίνεται κατάχραση του κανόνα σε ορισμένα κράτη-μέλη. ε, ε θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την Κομισιόν το εξή. Υπάρχει δυνατότητα να αναθεωρηθεί αυτός ο κανόνας ε, που εισήχθη ως ε, εξαίρεση για κάποια πολύ συγκεκριμένη και ειδική περίπτωση και τελικά έχει γενικευθεί από τη χρήση του από τις επιχειρήσεις με τρόπο διαφορετικό από αυτό που είχαμε προβλέψει. Δεύτερον, να ρωτήσω την Κομισιόν, σκέφτεται σε ό,τι αφορά το έλλειμμα εφαρμογής ε, για τον χρόνο ξεκούραση και την βραδινή οδήγηση θα έχει σκεφτεί ε, το θέμα των weekend bands, ε, δηλαδή αυτών των, ε, των, των απαγορεύσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, ε, μήπως θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. τρίτον, αστυνομική συνεργασία με την εφαρμογή της Νέας Συνδίκης Λισαβόνας. Είναι είναι δυνατόν να είμαστε πιο θετικοί σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ε, αστυνομικής ε, συνεργασίας ε, για την δίωξη των παραβάσεων. Voorzitter, dank. Dit is een onderwerp waar we eigenlijk veel langer over zouden moeten praten. En ik vind het dus jammer dat we zo. Ευχαριστώ είναι κρίμα που έχουμε τόσο λίγο χρόνο, λέει ο κ. Βαντάλεν. θα έπρεπε να έχουμε λίγο περισσότερες ευκαιρίες να μιλήσουμε. Μακάρι να είχαμε ε, το ίδιο σύστημα το Βλαδιβοστόκο κόστο Σάνον. Το πρόβλημα όμως είναι η, συμμόρφωση. Ε, με, οργανώσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο στις 22 Μαρτίου ε, μία ακρόαση παρουσία υψηλών στελεχών της Κομισιόν και εκεί κατάλαβα ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια νομοθεσία αλλά η συμμόρφωση με την νομοθεσία. Αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της ε, αυτό ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ο σεβασμός γιατί δεν διαθέτουμε ένα εγχειρίδιο ενιαίο που να εξηγεί πώς θα εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ε, ε, διατάξης νομοθεσίας. Δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία. Χρειαζόμαστε ένα εγχειρίδιο ενιαίο για να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες από το Γιβραρτάρ μέχρι τα σύνορα με την Πολωνία και την Ρωσία, από τη Φιλανδία μέχρι την Ελλάδα, έτσι ώστε ο καθένας να γνωρίζει ποιοι ακριβώς είναι οι κανόνες και πώς μπορεί να τους στηρίσει. Γιατί τίθανται πολλά ζητήματα Ερμηνεία των κανόνων. Συνεπώ, παρακαλώ μην αγγίξετε, μην αλλάξετε το νομοθετικό πλαίσιο. Ε, θα πρέπει να δραστηριοθούμε επί της εφαρμογής. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Το πρόβλημα επίσης, το άλλο πρόβλημα επίσης αφορά τους αυτοαπασχολούμενους δεν είναι δυνατόν το κράτος να παρεμβαίνει στην προσωπική τους ε, ζωή, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Μετρούμε το χρόνο που πηγαίνουν να κάνουν ψώνια, για παράδειγμα. Ε, γίνεται, γίνονται τρομακτικά λάθη και μετά από χρόνια τα παίρνει πίσω η Κομισιόν και λέει «Α, ναι, ναι, έχετε δίκιο, ήταν γελία». Ε, πρέπει να το πούμε. Ε, ας πούμε, η Ευρώπη έκανε ένα λάθος και ε, ας διορθώσει. Είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να διατηρηθεί αυτή η νομοθεσία για τους ε, αυτοπασχολούμενους. Είναι γελία. Είναι γελία. Είναι δηλαδή άνω ποταμών. Θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των αυτοαπασχολούμενων. Και όπως σας είπα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σεβασμό της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Στέρξ. Ε, Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Πέτερ μόλις τώρα. Είναι ήδη δύσκολο να γίνει σεβαστός ο χρόνος οδήγησης και ο χρόνος ξεκούρασης. Θα προτιμούσα να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Έχουμε φορτηγά και οχήματα που έχουν σταματήσει, σταματάνε τακτικά στη λωρίδα εκτεξανάγκης για ξεκούραση, αναγκαστική ξεκούραση και δημιουργούν πολλά προβλήματα ασφάλειας, για παράδειγμα. Συνεπώ η νομοθεσία είναι ήδη περίπλοκη. Αν τώρα κάνουμε και το λάθος να πούμε ότι θα ελέγχουμε έναν αυτοπασχολούμενο εκτός των ορών ε, εργασίας του ή ε, οδήγησης, κάτι που είναι και αδύνατο κατά βάση, ε, προσθέτουμε βάρος ακόμα μεγαλύτερο ε, σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Συνεπώς, διαφωνώ με τον έλεγχο των αυτοπασχολούμενων διότι με αυτόν τον τρόπο παρεμβαίνουμε στην προσωπική του ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτό το δικαίωμα να το κάνει. Εμεί ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να διορθώσουμε αυτό το μεγάλο σφάλμα. Μα λένε ε, για το ε, ισότητα για όλου. Ναι για το χρόνο εργασία και ναι για το χρόνο ξεκούραση. Αλλά αν ένα οδηγό θέλει να πάει να χορέψει το, το βράδυ, δεν είναι τον, να τον ελέγχουμε ε, αν είναι κουρασμένος Δευτέρα το πρωί, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να το δει με τον ειδικό τον εργοδότη. Λοιπόν, θα πρέπει να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Ίσως αυτό το λάθος, ε, ίσως δεν το έκανε η Κομισιόν, αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να το διορθώσει. Ε, ευχαριστώ κύριο ε, Σίλβα και ο συνάδελφός της Κομισιόν θα πρέπει να είμαι αυστηρός μαζί σας, ε, φοβούμαι, λέει ο Πρόεδρος, γιατί έχουμε μείνει πίσω και είχαμε Έχουμε μείνει 20 λεπτά πίσω και είχαμε μακροσκελείς τοποθετήσεις. Παρακαλώ, ο κύριος Σίλβα, για την εφαρμογή, πρόεδρε, δύο θύματα απλώ. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους. Η Γενική Οδηγία Χρονοεργασίας δεν αφορά, δεν εφαρμόζεται για τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτό είναι σαφές. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πράγματι υπάρχει ανάγκη απλούστευσης και ευελιξία των κανόνων και μερικές από τις επιλογές που προτείναμε στους κοινωνικού εταίρους εντός του πλαισίου ευρύτερα ήταν κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποίησεις προς καλύτερη ευελιξία. Δηλαδή η διεύρυνση της περίοδου αναφοράς για το χρόνο εργασίας εβδομαδιαίως Ωστόσο, δεν, να, ας μην ξεχνούμε ότι είναι οδηγία ασφάλειας στην εργασία και αυτό δεν αφορά το αν εργάζονται οι εργαζόμενοι σε μεγάλη ή μικρή επιχείρηση, ως προς την ασφάλεια δηλαδή. Ωστόσο, το εξετάσαμε το θέμα και περιμένουμε και την, ε, το input των ε, κοινωνικών εταίρων. για τις ε, μεταφορές ε, ή τους οδηγούς ε, για αποστάσεις μικρότερες των 50 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν ταχύγραφοι εδώ. Εδώ καλυπτόμαστε από την Γενική Οδηγία Χρόνου Εργασίας. Και το πρόβλημα είναι ότι η οδηγία αυτή ποσοτικοποιεί τους χρόνους ανάπαυσης, για παράδειγμα. Αλλά εκτός από τους εργαζομένους αυτούς συγκεκριμένα για τους χρόνους ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, για παράδειγμα. Και τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία με πολύ μεγάλο περιθώριο ευελιξίας. Σε κάποια κράτη-μέλη, λοιπόν, όπως ακούμε, δεν υπάρχει επαρκής προστασία των εργαζομένων αυτών. Για τις αστικές μεταφορές, για παράδειγμα. Συχνά έχουμε 6, 7, 8 ώρες συνεχούς υπηρεσία για τους οδηγούς χωρίς, επαρκή, χωρίς χρόνο ανάπαυσης διερευνούμε μερικές από τις περιπτώσεις αυτές και δεν έχουμε καθορίσει ακόμα μια σαφή παραβίαση. Απλώς έχουμε εκρεμίσει ακόμα υποθέσεις, παραμένουν ανοιχτές, δεν είναι θέμα μη εφαρμογής, είναι θέμα του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη τους κανόνες που δεν έχουν ποσοτικοποιημένες παραμέτρους για τις νυχτερινές βάρδιες ή τους χρόνους της περίοδους ανάπαυσης. Εν πάση έχουμε διαρευνήσει, δεν έχουμε διαδικασία παραβίαση αυτή τη στιγμή ανοιχτή. Να σα πω. Ο κύριο Πασκουαρέλη. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πάρα πολύ σύντομο και να ζητήσω από τα μέλη που δεν έχουν λάβει απάντηση από μένα να μας απευθύνουν οποιαδήποτε πρόσθετη ερώτηση είμαστε στη διάθεσή σα. Για τα θέματα επιβολή και εναρμόνιση των διαδικασιών παραβίαση, αυτό είχε τεθεί από πολλά μέλη, δεν θα ήθελα να εμείνουμε ιδιαίτερα στο θέμα της εφαρμογής. Η κατανόηση των, κανόνων είναι, ευρύτερα μιλώντας, η ίδια. Και υπάρχει μια συνεχή συμβολή σε μια κοινή ερμηνεία και κοινή κατανόηση των κατώνων. Όπως και χθε ακόμα είχαμε την ε, άποψη της ε, Ειδικής Επιτροπής για την ειδική εφαρμογή των κανόνων ε, χρόνων οδήγησης και χρόνων ανάπαυσης κτλ. Δουλεύουμε υπό τον περιορισμό των προηγούμενων συνθήκων βεβαίως. Παρά τα αυτά έχουμε εισαγάγει κανόνες για την κατηγοριοποίηση των παραβιάσεων και την αξιολόγησή του σύμφωνα με κάποια μια σειρά κριτηρίων ως προς τη σοβαρότητα της παραβίασης και όπως έλεγε και ο κύριος ε, Κράμερ για την βάση δεδομένων έχουμε την ERU, την ERU βάση δεδομένων που έχει οικοδομηθεί ακριβώς στο πλαίσιο της εφαρμογής του λεγόμενου road package το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται. Έχουμε αιτήσεις εκθέσεις και όταν τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τις ε, υποχρεώσεις τους, είτε τις απλές ε, υποχρεώσεις εκθέσεως, υποβολής εκθέσεως ή μη σωστής εφαρμογή, τότε έχουμε διαδικασίες παραβίασης, οι οποίες δημοσιοποιούνται. Έχουμε ανακοινώσει τύπου κάθε φορά που εκινούμε μια τέτοια διαδικασία. Το άλλο σημείο αφορούσε την υπερβολική γραφειοκρατία, τους ε, πρόσθετους κανόνες ε, και το γεγονός ότι η οδηγία χρόνου εργασίας έχει προεκταθεί να καλύπτει και τους αυτοαποσχολούμενους. Να σας θυμίσω εδώ ότι η Κομισιόν είχε προτείνει να διατηρηθεί η εξαίρεση των αυτοαποσχολούμενων από την οδηγία χρόνου εργασίας και το Κοινοβούλιο ήθελε να τη συμπεριλάβουμε μην μας κατηγορείτε λοιπόν σας παρακαλώ ότι εμείς προσθέτουμε στο νομοθετικό άκθος. Προσπαθούσαμε να αποφύγουμε εμείς να δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο τους κανόνες. Απλώς ζητήσαμε οι κανόνες υφιστάμενοι να εφαρμόζονται ορθώς, το οποίο είναι ευθύνη των κρατών μελών. Και εμείς θέλουμε το καλύτερο δυνατό μέλλον και την καλύτερη δυνατή ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις, αλλά με δίκαιου κανόνες ανταγωνισμού και δίκαιου κανόνες για την ασφάλεια των εργαζομένων. Εάν δεν έχουμε κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία επί της κοινωνικής διάστασης, τότε θα είχαμε 27 διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Αλληλοαντικρουόμενε. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του να έχουμε εναρμονισμένους κανόνε Και να θυμίσω στην Επιτροπή σα ότι βεβαίω μπορεί κανεί να αμφισβητεί τα μεγέθη, αλλά ο ψηφιακός ταχυγράφος έχει μειώσει το διοικητικό κόστος σε ένα μέγεθος 500 200 εκατομμύριων ευρώ, λοιπόν, η μείωση του διοικητικού κόστους. Εμείς έχουμε διενεργήσει αρκετές, ε, αρκετές πιλωτικά προγράμματα που έχουν οδηγήσει στην ε, σύσταση, αν θέλετε, στη δημιουργία όρων αναφοράς για ασφαλείς χώρους σταθμεύσεως. Έχουμε συγχρηματοδοτήσει αρκετές ε, πιλωτικές λοιπόν δραστηριότητες σχετικά με αυτό. Και είμαι στη διάθεσή σας και για αρκετά άλλα ερωτήματα, αλλά μας πιέζει ο χρόνος όπως είχατε πει και εσείς Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Καταρχήν, έχετε απρόλυτο δίκιο ότι το Κοινοβούλιο είχε επιμείνει για τους αυτοαπασχολούμενους και σωστά το έπραξε. Και δεύτερον, όσον αφορά τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης, ε, είμαι υπέρ των ασφαλών χώρων στάθμευσης, απλούστατα ε, πρέπει να πείσουμε αυτούς ε, οι οποίοι ζουν δίπλα σε αυτούς τους χώρους γιατί κανείς δεν το θέλει πίσω από το σπίτι του τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο Σας ευχαριστώ και όσον αφορά το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Φλέκενστάιν για την ΕΜΣΑ. Κύριε Φλέκενστάιν έχετε το λόγο και αν... Ε, ε, ε, ε μου επιτρέψετε θα αποχωρήσω για δύο λεπτά και επανέρχομαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε εκφράσει επανειλημμένως την ικανοποίησή μας ε, για την εργασία αυτή και μέχρι σήμερα ε, ο βασικός κανονισμός επί του θέματος έχει αλλάξει και ε, θα έπρεπε τώρα να το εξετάσουμε κάπως πιο μακροπρόθεσμα. Η ε, πρόταση της ε, Επιτροπής είναι να διευκρινίσουμε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΜΣΑ και τους τομείς στους οποίους εστιάζεται. Η επεξεργασία της πρότασης αυτής λοιπόν βασίζεται εις μία συνεννόηση των επι των υπευθύνων για την ΕΜΣΑ το 2008, μία αξιολόγηση της ΕΜΣΑ, ε, μία επιπλέον αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων για την ΕΜΣΑ του 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τέλος μία, μία σύσταση της ΕΜΣΑ όπου εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη ε, η οποία επακολούθησε. Νομίζω ότι ε, η ε, οργάνωση αυτή μπορεί να συμβάλλει και σε άλλα θέματα για την εποπτεία της ολοκληρωμένης θαλασσίας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί μπορεί να αναλύσει τις επιπτώσεις ε, των θαλασσίων μεταφορών εις ε, το περιβάλλον και ε, έχουμε χρησιμοποιήσει ούτως ή άλλως τις αξιολογήσεις του οργανισμού αυτού και μέχρι σήμερα ικανοποιητικά. Έχουμε δύο εκθέσεις του κυρίου Μπεγκράνης και πρόσφατα την έκθεση Rotman Call που αναφέρεται στη ρήπανση των θαλασσών και ε, το θέμα μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και πλοίων τα οποία μας απασχολούν και η έκθεση για την ολοκληρωμένη ε, Επιτροπή των Θαλασσών όπου ε, ζητούμε ε, να αναλάβει η ΕΜΣΑ την επιθεώρηση των υπερακτίων εγκαταστάσεων και η ΕΜΖΑ μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απεδέχθη η ΕΜΣΑ να αναλάβει αυτές τις, ε, ε, τις εγκαταστάσεις και τον έλεγχο τους ε, και να χρηματοδοτηθεί προς αυτή την κατεύθυνση διότι το Συμβούλιο όπως γνωρίζετε έχει μια πολύ περιοριστική στάση και οι συζητήσεις στο Συμβούλιο δεν είναι βίωνες σχετικά με μια διεύρυνση των καθηκόντων του οργανισμού αυτού. Αλλά πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σωστή σε πολλά σημεία και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά 4-5 θέματα. Καταρχήν όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση πετρελαιοκυλίδων νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε και μπορούμε να το πούμε εδώ ιδίως για τις πλατφόρμες πετρελαιοπαραγωγής. Βεβαίως πρέπει να εξετάσουμε γιατί δεν μπορεί κανείς αποτελεσματικά να διαλύσει αυτές τις κυλίδες και πέραν αυτού πώς μπορούμε να ασκήσουμε καλύτερη πρόληψη. Είναι κάτι που πρέπει να ξανασκεφτούμε. Δεύτερο θέμα. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο αυτό το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή την τεχνική συνεργασία με τις γειτονικές χώρες που πρέπει να βελτιωθεί, διότι αν υπάρχει μία τέτοια οικολογική καταστροφή από πετρέλαιο σε μια γειτονική χώρα όλοι πλήττονται, όλοι οι γείτονες. Και η Επιτροπή αυτή στηρίζει εδώ και χρόνια την ιδέα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού θαλασσίου χώρου όπου οι μεταφορές επιβατών και αγαθών δεν θα υπόκεινται σε πολλές διατυπώσεις και αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι επίσης αυτό να επιταθεί με την εμπλοκή της ΕΜΖΑ και εις ε, τις ε, τελωνιακές διαδικασίες αλλά και εις ε, την παρακολούθηση των διαφόρων μεθόδων μεταφοράς. Ε, και τέλος πιστεύουμε ότι θα είναι θετικό αν ε, η ΕΜΣΑ βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιθεώρηση ε, επί των πλοίων σε συνεργασία με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την επιθεώρηση και εποπτεία των λιμένων ε, και των εγκαταστάσεών τους. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και τέλος, ε, ε, δύο θέματα που με ενδιαφέρουν θα τονίσω κλείνοντας. Καταρχήν, αν η ΕΜΣΑ θα μπορούσε να συμβάλλει ή στην πιστοποίηση στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων τα οποία εμείς ε, ε, διατυπώνουμε σαν προτάσεις και δεύτερον για τα διπλώματα ε, ικανότητος των ναυτικών εάν δηλαδή η ΕΜΖΑ μπορεί να επισκεφθεί όλες τις ναυτικές σχολές οι οποίες υπάρχουν διεθνώς και να παρακολουθήσει αν το πρόγραμμά τους και τα πιστοποιητικά που εκδίδουν συνάδουν με την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει. Ιδίω εάν αναφερόμαστε εις ε, την εφαρμογή της ε, συμφωνίας για την εργασία στη θάλασσα. Ε, είχαμε μία πρώτη συζήτηση με, μεταξύ εισηγητού και σκιωδών εισηγητών ε, βεβαίως ε, η πολιτική ομάδα ECR έχει διαφορετική άποψη, η ε, Ευρωπαϊκή Συντηρητική δηλαδή, και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, διότι δεδομένη της στάσης του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή θα χρειαστούμε μια σαφή πλειοψηφία και γι' αυτό θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε σε ορισμένα θέματα κατά τρόπον ώστε και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν αλλά και από την άλλη πλευρά να δούμε ε, ρεαλιστικά τι θα μπορέσει να περάσει από το Συμβούλιο. Και γι' αυτό ε, θα ζητούσαμε από αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη πείρα να μας πούν πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Φραγκενστάιν. Εννιά ομιλητέ, αν μετράω καλά, παρακαλώ πολύ να είστε σύντομοι. Οι σκιώδεις εισηγητέ τρία λεπτά, οι υπόλοιποι δύο λεπτά. Ουφ, όλο και πιο μακροσκελής γίνεται ο κατάλογος. Κύριος Πασκουάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Φλάκεστάιν, όπως ε, είπε ε, ήταν πολύ ε, ήταν πολύ σοβαρός με όλους μας. Το έγγραφο εργασία που ετοίμασε ε, μπορεί να αποτελέσει βάση εργασία ε, για ένα συμβασμό. Είναι δύσκολη η κατάσταση, έχουμε οικονομικές δυσκολίες, το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ αυστηρό και θα ε, δημιουργήσει σημαντικά προσκόμματα στην ε, ε, χορήγηση νέων αρμοδιοτήτων στον ΕΜΣΑ. Τον Δεκέμβρη, όταν ο Ντερόιτερ, ο διευθυντής της υπηρεσίας αυτής, εμφανίστηκε ενώπιον μας, μας είπε ότι θα πρέπει το προσωπικό να αυξηθεί κατά 18 άτομα, 3,9 εκατομμύρια ευρώ αυξητού προϋπολογισμού. Ε, αυτό μας τρόμαξε. Θα πρέπει να, ε, να βρούμε μια λύση. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ε, υπάρχουν θέματα στα οποία το Συμβούλιο ε, είναι υπερβολικό. Ε, ε, μας ε, ζητούν ε, χρήση επιτροπολογίας. Ε, διαφωνεί το Συμβούλιο με τις προτάσεις για τους ελεγκτές στα κράτη-μέλη. Δεν θέλουν ε, καινούργιες αρμοδιότητες στο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλής Θάλασσας. σε αυτό το θέμα. Επίσης το Συμβούλιο θέτει το θέμα των πόρων της χρηματοδότησης. Ε, μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση, εντάξει, δεν ε, υπάρχει ε, λόγος να φτάσουμε στα άκρα. Νομίζω ότι το Συμβούλιο μπορεί να δράσει εξισορροπητικά. το, η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει πολύ γρήγορα, η, το Συμβούλιο καθυστερεί, και δημιουργεί προσκόμματα, εμείς μπορούμε να ε, παίξουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι ε, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Θάλασσα ω τώρα έχει παίξει ένα πολύ καλό ρόλο και νομίζω ότι είναι χρήσιμος. Ε, τώρα, το κατά πόσον ο ΕΜΣΑ πρέπει να αναλάβει αρμοδιότητες ορισμένε από τι αρμόδιε που αναφέρεται το έγγραφο έχω κάποιε αμφιβολίε. Σε ό,τι αφορά τι πιστοποιήσει, αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Ήδη στο, ε, στο παρελθόν ε, είχαμε προβλήματα με την αμοιβή αναγνώριση. Τώρα μιλάμε και για πιστοποίηση. Ε, είναι, είναι αδύνατον. Μετά, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Δανία δεν συμφωνούν με το, με το, με τις, ε, το θέμα των εξέδρων τη πετρελαίου και φυσικού αερίου υπεράκτια ε, και τον έλεγχο από τον ΕΜΣΑ. Ε, Κοιτάξτε τι έγινε στο, Μεξικό. Το, η, η εξέδρα στο, στο κόλπο του Μεξικό ε, ήταν εκτός ελέγχου και είδατε ποιο είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την ε, μόλυνση από Ε, οι σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον και ο δόλος θα πρέπει να τιμωρούνται. Ε, δεν θα αργήσω, Πρόεδρε, δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα, να επαναλάβω μόνο το εξή ότι ο δρόμος είναι ο δρόμος ε, του εισηγητή. Να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε μια ισορροπημένη θέση του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να διευκολύνουμε το έργο της Κομισιόν και ταυτόχρονα ε, να καταρρίψουμε αυτή την πολύ αυστηρή και αρνητική θέση του Συμβουλίου. Α μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι γιατί δεν θα πετύχουμε τίποτα. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φλακεστάιν για την ε, μεθοδολογία του, μεθοδολογία που έχει ακολουθήσει. Η, η, η, ε, ο, ο οργανισμός δημιουργήθηκε μετά την κρίση του Έρικα και την συνεπακολουθή Το 2003, μάλλον από το 2003 και μετά, έχει τροποποιηθεί σε ε, τρεις περιπτώσεις. Ε, πρώτον, μετά την κρίση του πρεστής. Οπότε στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ορίσουμε καλύτερα την αποστολή του ΕΜΣΑ. Έχει γίνει εξωτερική αξιολόγηση, έχει γίνει αξιολόγηση πλευρά της Κομισιόν, έχουμε τις ε, καινούριε αρμοδιότητες μέσω τρίτου πακέτου ασφάλειας θάλασσα. Έχουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2010 όπου ζητείται να συμπεριληφθούν και εγκαταστάσεις, οι υπεράκτες εγκαταστάσεις άντλησης και συνεπώς η Επιτροπή ε, εργάζεται εδώ και αρκετό ε, καιρό για τον ενίο θαλάσσιο χώρο στην Ευρώπη Οπότε η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του, του ΕΜΣΑ θα πήγαινε προ αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε έχει ζητήσει επανειλημμένως το Κοινοβούλιο τέτοιε αλλαγέ, ε, συνεπώ θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε τώρα. Τώρα, τι σημαίνει η διεύρυνση αρμοδιοτήτων του ΕΜΣΑ. Συμφωνώ με τον ρόλο της κατάρτισης και της ε, πιστοποίηση δικτύου ακαδημιών. Είναι πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μια ε, σχολή κατάρτισης ε, ε, διεθνούς εμβέλειας. Είναι πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, είναι πολύ σημαντική η συμπερίληψη των εγκαταστάσεων άντλησης και τη δυνατότητα ο ΕΜΣΑ να χορέγει τα πιστοποιητικά. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν στην οικοδόμηση αυτού του ενιαίου θαλάσσιου χώρου στην Ευρώπη, που θα είναι ενιαίος, εναρμονισμένος, αποτελεσματικός και αποδοτικός. Θα μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές κρίσεις. Δεν πρέπει οι τροποποιήσεις κάθε φορά να έρχονται μετά από μια κρίση. Ο ΕΜΣΑ δεν είναι δυνατόν να οικοδομείται ε, μόνο ε, όταν το επιτάσσουν τα γεγονότα. Πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να αναλύσουμε τις συνέπειες όχι μόνο της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής αλλά και της συνέπειας της ένταξης των διαφορετικών σχολών στη δημιουργία ενό ενός δικτύου ή στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σχολής. Θα πρέπει να αναλύσουμε τι έχει το κάθε κράτος μέρος, τι διαθέτει, τι μπορεί να συνεισφέρει και όλα αυτά να τα ενοποιήσουμε. Συμφωνώ με την θέση του κ. Ντεγκράντες. Θα πρέπει να καταλήξουμε μια συμφωνία, αλλά κα, ε, κατά την μου πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, γιατί θα πρέπει να στοιχηματίσουμε υπέρ ε, ευρωπαϊκών project, υπέρ της ευρωπαϊκής προσέγγισης, γιατί τα κράτη-μέλη επιθυμούν απλώς να διατηρήσουν τις αρμόδιες τους και αυτό θα πλήξει το μέλλον. Mr. Taylor. Uh, thanks, Chair. Κύριε Στέιλο, ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς γενικά υποστηρίζουμε και την κατεύθυνση του εγγράφου εργασία του κυρίου Φλάκενστάιν αλλά και την ε, προέκταση του πεδίου της ΕΜΣΑ στο πεδίο όπου δεν θα υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με το έργο άλλων οργανισμών. Αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι θα πρέπει οι υποχρεώσεις που έχει η ΕΜΣΑ να συνοδεύεται και από τους απαραίτητους πόρους και τα μέσα που θα πρέπει να έχει η διάθεσή της. Τώρα για τις προτεραιότητες της εργασίας που ε, θα επιλεγεί θα πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον από τις επιχειρήσεις άντλησης ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ε, ε, ήμασταν υπέρ και των ελέγχων λιμένος ε, και την, ε, τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών και την περιβαλλοντική περιβαλλοντικά ορθή συμπεριφορά, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις περιβαλλοντικές αποδόσεις των επιχειρήσεων δεν έχουμε επαρκή δεδομένα. Έχουμε λυπή δεδομένα θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα επίσης βελτιωμένο παρακολούθησης ε, των σκαφών, ιδιαίτερα αυτών που ε, έχουν ε, επικίνδυνα φορτία, για την επέκταση και του καλύτερη, της καλύτερης λειτουργίας του Net Επίσης θα πρέπει να έχουμε έναν ανεξάρτητο οργανισμό που να ελέγχει καλύτερα τις, ε, τα σκάφη όπως και τα πληρώματα για την ασφάλεια των μεταφορών. Ευχαριστώ κύριος Βαντάμ, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το έργο της ΕΜΣΑ είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι από τους οργανισμούς που καλύτερα λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω δύο φορές. Τώρα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά λέμε ότι πρέπει να κάνουμε όλο ένα και περισσότερα, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη κτλ. Αλλά δεν διαρωτώμαθα κατά πόσον πράγματι όλα αυτά που ζητούμε είναι απαραίτητα ή μήπως η φυστάμενη κατάσταση είναι επαρκής, το πλαίσιο είναι επαρκής και απλώς χρειάζεται να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και συχνά δεν είναι μόνο θέμα αποτελεσματικότητας, λέγεται, αλλά χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη και τότε όλα θα πάνε καλά. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η τάση, αυτό το όρομα δεν είναι πάρα πολύ μακρόπνο αν θέλετε. Δεν βλέπει πολύ μακριά. Δεν είναι απαραίτητο να εισαγάγουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες ε, για την έμψα για την, ειδικά σε ό,τι αναφορά την εσωτερική πλοήγηση. Γιατί δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά. Έχουμε ήδη μια επιτροπή στο Στρασβούργο που λειτουργεί άριστα πολλά πολλά χρόνια τώρα και θα συνεχίσει να το κάνει σε στενή συνεργασία με την Joint Working Group Επομένω, δεν είμαστε στο πεδίο της συζήτηση των αρμοδιοτήτων της ΕΜΣΑ. Για του ελεγχού λιμένους και εδώ έχουμε ε, οργανισμό, αρχή που λειτουργεί εξαιρετικά και έχουμε και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και άλλα κράτη Ούτε αυτό λοιπόν χρειάζεται να το υποβάλουμε, να το εισαγάγουμε στις αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ γιατί θα αποφύγουμε περιπλοκές και ασάφεια. Έχουμε οργανισμούς και βήματα που λειτουργούν ωραιότατα αυτή τη στιγμή. Όπως αυτό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των σχετικών σχολών, ούτε αυτό χρειάζεται να το εισαγάγουμε στις αρμοδιότητες της ΕΜΣΑ. Η, Άννα, η απόφυτη επιθυμούν να συνεχίσουν μέσα στην ευσυπλοεία και υπάρχουν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα υποβάλουμε στο πλαίσιο της ΕΜΣΑ. Δεν έχει νόημα. Πρόεδρε, ο εισηγητής ήδη μας είπε, ήδη μας ανέφερε ότι ασκούνται έντονες κριτικές και εγώ εκπλήσωμαι πρέπει να σας πω σχετικά με το πώς προχωρούμε. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να τονίζουμε και ξανατονίζουμε να επικαλούμε θα την περισσότερη Ευρώπη. Η ΕΜΣΑ μια χαρά λειτουργία παραλαμβάνω. Μπορούμε απλώς και θα έπρεπε να διέπουμε καλύτερα τις αρμοδιότητες που έχουμε και όχι να προσθέτουμε. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομα. Βεβαίως, πολύ θα ήθελα να, υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό μπορεί να γίνει με τα, ε, μέσω διαφόρων οργανισμών αλλά καταρχήν εδώ μιλάμε για έναν οργανισμό ασφαλείας ε, και όχι για άλλα θέματα. Δεύτερον, η επέκταση των ε, ευθυνών αλλάζει τη φύση του οργανισμού και δεν ενισχύει τις αρμοδιότητες στα θέματα των, ε, της ασφαλείας αντιθέτως την αποδυναμώνει διότι προτείνουμε να καλύψει ασαφείς τομείς το η ηλεκτρονική ναυτιλία, την νομοθεσία, συστήματα δηλαδή που δεν ελέγχονται πλήρως και που διηλίζουν τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Δεύτερον υπάρχουν επιφυλάξεις διότι υπάρχουν προτάσεις οι οποίες είναι αντίθετες με τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών όπως ο έλεγχος των λιμανιών και ούτω καθεξής. Και τρίτον, όσον αφορά τις υπερπόντιες πλατφόρμες αντλήσεως πετρελαίου, ε, νομίζω ότι ε, μη ένας οργανισμός ασφαλείας μπορεί να ελέγξει αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι ε, και ορυχεία πλέον των ναυτικών οικοδομημάτων και δεν καλύπτεται από τη, η εντολή του οργανισμού από αυτή την περιγραφή. Οπότε πιστεύω ότι εάν ε, αν θέλει κανείς να συμμετάσχει εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλους διεθνείς οργανισμούς με αυτή την οργάνωση δεν είναι σωστό. θα, αν αλλάξουμε την διάταξη θα πρέπει να αλλάξουμε και τους πόρους χρηματοδότησης γιατί αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή ε, ε, οργάνωση ε, δεν πρέπει να οδηγήσει σε μία παραμόρφωση αυτού του οργανισμού που θα μειώσει την αποτελεσματικότητά του. Ε, ε, η κυρία Μάισνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ τόση ώρα διότι μου αρέσει αυτή η έκθεση και καλύπτει πολλά θέματα που είπαμε αλλού και έτσι τώρα θα αναφερθώ μόνο σε δύο θέματα που μου φαίνονται σημαντικά ε, δηλαδή όσον αφορά την αρμοδιότητα της ΕΜΖΑ και την ακτοφυλακή. Είναι δύο θέματα σε τα οποία θεωρώ θετικά Τώρα, πώ θα συνεννοηθούμε και θα συντονιστούμε είναι κάτι που θα δούμε, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φλέγκενστάιν για την εργασία την οποία ε, έχει καταρτήσει. Ευχαριστώ η κυρία Φώστερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Συμφωνώ με ορισμένους συναδέλφους, τον κύριο Βαντάλεν και τον κύριο Ρικέ. Ε, δηλαδή δεν πρέπει να αποκλίνουμε από το ρόλο που πρέπει να καλύψει η ΕΜΣΑ διότι όταν ε, μιλάμε, μιλήσαμε για τη ε, δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας ε, ώρες ώρες προτρέχουμε των εξελίξεων ε, και δεν ε, αυξάνει κανείς την αποτελεσματικότητα ή μειώνει το κόστος ε, υπάρχουν επικαλύψεις και χάνει την κατεύθυνση την οποία επιζητεί Γι' αυτό και θεωρώ ότι η ΕΜΣΑ κάνει εξαιρετική εργασία για πολύ σωστούς λόγους. Αλλά όσον αφορά α, το, τις αρμοδιότητές της είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Επίσης αναφέρθηκαμε στις εγκαταστάσεις αντλήσεως πετρελαίου και αερίου και δεν νομίζω ότι εκεί έχει αρμοδιότητα ή θα έπρεπε να έχει αρμοδιότητα η ΕΜΣΑ ε, σε τέτοιες, οργαν... σε τέτοιες εγκαταστάσεις διότι εφόσον συνάδουν με τις διεθνείς συμβάσεις όλας και ε, όσον αφορά τις υποδομές τους πρέπει να είμαστε ε, αισιόδοξοι. Δηλαδή νομίζω ότι έχουμε πολύ υψηλές προδιαγραφές για τις ε, εγκαταστάσεις, τις πλατφόρμες οι οποίες οποίες ε, ε, βρίσκονται ε, πέραν των ακτών για την άντληση πετρελαίου και δεν θα συμφωνούσαμε την στήριξη της ΕΜΖΑ σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι ε, υπάρχουν θέματα που θα συμφωνούσα. Τέλος, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, όλα καταλήγουν στη χρηματοδότηση και οποιαδήποτε ε, οποιαδήποτε χρηματοδότηση θα πρέπει να αυξηθεί ε, εις βάρος κάποιας άλλης, κάποιο άλλο κεφαλαίο και γι' αυτό πρέπει να, να το προσέξουμε. Ο κύριος Κιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Φλέκενστάιν και τον κύριο Ντεγκράντερ, όλους τους εισηγητές και όντως είδαμε ότι στον τομέα της ασφαλεία, ναυτικής ασφαλείας όσον αφορά τους ελέγχους έχουμε ε, διάφορους τέτοιους ελέγχους ιδίως σε εθνικό επίπεδο ε, και είτε μέσω εθνικών συστημάτων ή μέσω του IMO ε, υπάρχει εφαρμογή διαφόρων κώδικων, μαρπόλ και ούτω καθεξής όλα αυτά εφαρμόζονται. Και αυτό ε, όταν όμως μιλάμε για ευρωπαϊκά ύδατα τότε οι αρχές ε, ε, θέλουν να ελέγξουν τις αρμοδιότητες και στην περίπτωση αυτή είναι εθνικού επίπεδου και το είδαμε και στην περίπτωση του ατυχήματος του Έρικα. Το ίδιο έχουμε και για τα φορτηγά. Υπάρχουν και διεθνείς οργανώσεις και εθνικές οργανώσεις και πάντοτε όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό επίπεδο μετακυλούμε την ευθύνη στην Ευρώπη χωρίς να υπάρχει εκτελεστικός οργανισμός. Τα κράτη-μέλη πρέπει να σκεφτούν τι αποθέματα έχουν στις εθνικές αρχές τους όσον αφορά την ακτοφυλακή παραδείγματος χάρη ή ε, το τελωνίο διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ε, ε, κάποιο αρμόδιο πλοίο το ίδιο και για την αλία κάποιο εθνικό πλοίο έρχεται και ελέγχει δεν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι ε, θα πρέπει να δούμε πως μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και τις ανταλλαγές και το συντονισμό γιατί έχουμε μία δυνατότητα να προβάλλουμε διάφορα θέματα και πρέπει να το συζητήσουμε το Συμβούλιο και να δούμε πώς θα το επιλύσουμε. Ευχαριστώ. Πριν μιλήσει ο κύριος Καραμίτσος, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που έθιξε ο κύριος Κιούν. Ε, θυμάμαι το Πρεστίζ, ήμουνα στην Επιτροπή Έρευνας του Prestige και εκεί ελέγχθη ότι ήταν λάθος των κρατών μελών. Για το Έρικα επίσης. Όταν βυθίστηκε το Έρικα ένας Γάλλος πρόεδρος είπε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ευρωπαϊκή δράση και ε, αυτά ήταν ήδη συμπεφωνημένα. Οπότε δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά, ζητάμε από την Ευρώπη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να αναλάβει την προσπάθεια, να επέμβει κτλ. Και όταν ε, θα πρέπει να προχωρήσει κανείς στην εφαρμογή, τα κράτη αρνούνται να συνεργαστούν. Οπότε δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να πρέπει να τα κάνει όλα, ούτε ότι όλα πρέπει να αναλαμβάνονται από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένοι σε ένα κόμμα και άλλοι σε άλλο. Ο κύριος Καραμίτσος έχει το λόγο. Με καλύψατε πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι σαφές για αυτούς από εμά που ήμασταν εκεί στις έρευνες ε, των Πρεστίζ και Έρικα, είχε γίνει πολύ δουλειά Κανένας δεν απορρίπτει την ιδέα ότι ήταν πολύ χρήσιμη εμπειρία, ε, ε, βάση περιπτώσει, ότι η συνεισφορά που είχαμε από την ΕΜΣΑ ήταν πολύ χρήσιμη. Αλλά να θυμίσω ότι όταν συζητούσαμε το τρίτο πακέτο ασφάλειας, υπήρχαν αρκετές ε, προτάσεις να βάλουμε συγκεκριμένα πράγματα στην αρμοδιότητα της ΕΜΣΑ και είχαμε ε, αποφασίσει στο τέλος της διαδικασίας ότι αυτό δεν ήταν κατάλληλο και θα προσαρμόζαμε τον κανονισμό ΕΜΣΑ στην επόμενη φάση όταν θα το ενισχύ το πακέτο. Είχαμε τις ε, έρευνες ατυχημάτων. Αυτό έγινε και τότε και το κάναμε και τώρα. Το άλλο που ήθελα να θυμίσω είναι ότι η πρόταση αυτή βασίζεται όχι μόνο στην εμπειρία που είχαμε και αυτό και στις απαιτήσεις του τρίτου πακέτου, αλλά και στις συστάσεις του προέδριου και στις εξωτερικές αξιολογήσεις που είχε δεχθεί το ίδιο το Προεδρείο. Αυτό που κάναμε στην πρόταση ήταν δύο στην ουσία πράγματα. Το ένα αφορούσε τη διακυβέρνηση. Είχαμε πει ότι οι μικρέ τροποποιήσει ε, για την διακυβέρνηση του οργανισμού για να αποφύγουμε σύγκρουση συμφερόντων με τα μέλη του Προεδρείου ήταν κάτι πολύ απλό. Εξού και η επιτροπολογία, κάτι που γινόταν ήδη με την ΕΑΣΑ. Και επίση είχαμε ζητήσει από τον διοικητικό διευθυντή να μην έχει την αρμοδιότητα μόνο αυτός, αλλά να υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα και από πλευρά σκάφους, αν θέλετε. Επιχειρήσαμε κάποια εναρμόνιση των στοιχείων αυτών μεταξύ των υπολείπων οργανισμών, πώς θα πρέπει να εκλέγονται οι διευθυντές κτλ. Πάντως, μείναμε σε σχέση με το πακέτο στην ίδια γραμμή προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας. Δεν είχαμε πει δηλαδή σε καμιά περίπτωση ότι θα διαβρύνουμε το πεδίο ή ότι θα το κατακαιρματίσουμε. Ωστόσο, είχαμε, έχουμε μάλλον αναπτύξει την εμπειρογνωμοσύνη, έχουμε πράγματα να κάνουμε, δεν θα ήταν ευφυές να δημιουργήσουμε ένα εξωτερικό φορέα που ήδη ο οργανισμός μπορεί να κάνει με προστιθέμενη αξία. Και αυτό είναι και το θέμα του Blue Belt, όπως λέγεται, της παρακολούθησης και των ελέγχων της ε, οδηγίας ε, διευκόλυνσης άλλο ένα θέμα ώστε να έχουμε αυτό το κοινό θαλάσσιο χώρο και να χρησιμοποιούμε τα μέσα και την εμπειρογνωμοσύνη 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε τη δυνατότητα και επομένως το να πάμε ε, σε εξωτερικό φορέα, στα ηλεκτρονικά τελωνία ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήταν ευφυές. Ας χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε μας και στην ΕΜΣΑ και να, ας τα χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Υπάρχουν τώρα κάποια άλλα θέματα για το e-maritime, και τις ε, εσωτερικές ε, υδάτινες οδούς, εκεί δεν πρέπει να έχουμε νέο οργανισμό. Εάν η ΕΜΣΑ ε, ελέγξει ε, μειολόγια, δεν θα ήταν... Δεν θα έπρεπε την ίδια στιγμή, χωρίς πρόσθετο κόστος, να τους ζητήσουμε να τους ελέγξουν πώς οι ίδιοι οργανισμοί που εργάζονται και στην εσωτερική, στις ιστορικές οδούς κάνουν τη δουλειά της. Το άλλο τώρα. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ του net και των υπηρεσιών πληροφοριών για τις ε, ποτάμιες οδούς. Γιατί αν χρειάζεται να έχουμε μια κίνηση μέσα στην ίδια ποτάμια οδό και περάσουμε από ένα διοικητικό σύστημα σε ένα άλλο διοικητικό σύστημα δεν θα ήταν πάρα πολύ πρακτικό. Αυτά είναι τα θέματα που συνδέονται με τις ε, εσωτερικές ε, οδούς. Ωστόσο δεν ήταν η πρόθεσή μας να προτείνουμε τη δημιουργία νέου οργανισμού υπεύθυνου για τις εσωτερικές ε, οδούς. Τώρα για τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου πρέπει καταρχάς να δούμε πώς οι εξέδρες αυτές πρέπει να ελέγχονται. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή και αυτό που είχαν κατανοήσει όλοι είναι ότι χρησιμοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε στη διαθέσή μας μετά από πιθανό ατύχημα. Δηλαδή, σε περίπτωση μόλυνσης, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα, τα σκάφη της ΕΜΣΑ για να καθαρίσουμε, για επιχειρήσεις ε, καθαρισμού και όχι για ελέγχους των εξέδρων, γιατί δεν έχουμε την, το νομοθετικό μέσο στη διάθεσή μας. Αυτά είναι μερικά από αυτά που ήθελα να πω, Πρόεδρε, και Σίγουρα θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και στο μέλλον να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ε, ο κύριος ε, Φλέκενστάιν θέλει κάτι να προσθέσει. Όχι κύριε Πρόεδρε. Όχι κύριε Πρόεδρε, σημείωσα όσα ελέγχθησαν, θα καταρτήσω την πρότασή μου, θα τη συζητήσω με τους κοιόδης συζητητές και θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 29 Ιουνίου, να ψηφιστεί στην Επιτροπή τον Οκτώβριο και να πάει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Και το τελευταίο θέμα που έχουμε προσυζήτηση είναι η Ευρωπαϊκή Οδική Ασφάλεια με εισηγητή τον κύριο Κόχ με συγχωρείτε για την προχωρημένη ώρα προσπάθησα να επαναφέρω στην τάξη τους συναδέλφους αλλά τώρα έχετε εσείς το λόγο Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Προτού προχωρήσω στις τροπολογίες θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, ε, τον πρόεδρο Σίμψον για το πρωινό εργασίας που είχαμε. Ε, συζητήσαμε πολλά θέματα. Σήμερα μπορώ να πω ότι όλα έχουν εξεταστεί και υποβάλλεται μία καλή έκθεση. Αναφερόμαστε εις το απρό τα προβλήματα των ε, τροχών, των ελαστικών, το, ε, της χρήσης ναρκωτικών ινοπνεύματος, στις ε, δυνατότητες προστασίας των παιδιών, στον οδικό κώδικα, όλα τα θέματα που θα καλύψει η έκθεση και τώρα έρχομαι στις τροπολογίες. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ε, κατέθεσαν τις 262 υπολογίες και ε, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες που ενισχύουν την έκθεσή μου και είναι η σωστή βάση για ένα πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πρόγραμμα που προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε. Ορισμένες τροπολογίες μπορώ να στηρίξω διότι είναι καινοτόμες, άλλες είναι ε, ε, πιο συγκεκριμένες και θα προβώ σε ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες θα συζητήσω ήδη την Πέμπτη με τους χειώδεις συζητές. Ορισμένες τροπολογίες άλλες θα απορρίψω. Παρακαλώ να έχετε κατανόηση διότι πιστεύω ότι δεν έχουν ε, σχέση με την ασφάλεια των οδικών μεταφορών αλλά με θέματα περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και άλλες τροπολογίες καλύπτονται ίσως από άλλες προτάσεις και ε, ε, ίσως ε, θα χρειαστεί επί ορισμένων θεμάτων να υπάρξει μία νέα οδηγία, ένας κανονισμός, ένα νέο πρόγραμμα και όσον αφορά τις τροπολογίες που μπορώ να αποδεχτώ αυτές προέρχονται από όλες τις πολιτικές ομάδες η κυρία Βίλς παραδείγματος χάρη προτείνει διάφορες λύσεις δηλαδή επάνδρωση με κάμερες του οδικού συστήματος και συμφωνώ ιδίως για θανατηφόρα ατυχήματα και ε, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να ε, απαντήσουμε στην πρόκληση η οποία δημιουργείται ε, από την στρατηγική για το 2020. Θέλω να τονίσω επίσης ότι όλες οι προσπάθειες δεν μπορούν να καταβληθούν μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λάβουν ε, τις ευθύνες τους και τα κράτη-μέλη. Ε, ε, επίσης μία άλλη τροπολογία η οποία αναφέρεται εις την χρήση ορισμένων ελαστικών για την, για την σωστότερη εφαρμογή θα πρέπει να στηριχθεί όπως άλλωστε και η τροπολογία που αναφέρεται στο δίπλωμα οδήγησης. Ε, ευχαριστώ επίσης ε, για την ε, επισήμανση για τα θανατηφόρα ατυχήματα σε διαβάσεις πεζών που είναι κάτι που θα τονίσω. Όσον αφορά την ε, ε, απαγόρευση οδηγήσεως υπό τη χρήση και την επίρρεια ναρκωτικών συμφωνώ αλλά επίσης ε, και η κόπωση επηρεάζει αρνητικά την οδήγηση και γι' αυτό χρειαζόμαστε μία ενιαία ρύθμιση για ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως σας είπα ορισμένες τροπολογίες θα τις απορρίψω όχι γιατί είναι λαθασμένες αλλά γιατί καλύπτονται σε άλλο κάποιο σημείο και απορριθμίζουν ε, τον ήρμο του, κειμένου. Ε, σε ε, ορισμένα σημεία θα ζητήσω να υπάρξει απόρριψη των τροπολογιών όπως παραδείγματο χάνει στην περίπτωση της τροπολογίας Μπασίτης όπου αναφέρεται οφείλεται εις ε, την ε, μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων που επλέκονται παιδιά καλύπτεται σε κάποιο άλλο σημείο επίσης για τους ποδηλάτες ε, καλύπτουμε το σημείο αυτό κάπου αλλού και υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες λίγες με τις οποίες δεν συμφορώ καθόλου δηλαδή να μειωθεί η ταχύτητα των μικρών φορτηγών διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχει μία μελέτη ότι δεν ε, η οποία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αυτά τα μικρά επαγγελματικά φορτηγά σε περίπτωση ατυχήματος. Όσον αφορά του εξωτερικά, τις εξωτερικές δαπάνες οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν, νομίζω ότι δεν μιλάμε εδώ για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των οδικών μεταφορών και ως εκ θα παρακαλούσα τον Ετούντα να αποσύρει την τροπολογία αυτά. Η κυρία Κρίσμπεκ ζητά η, η οδηγή των φορτηγών οδηγών να τιμωρούνται ιδιαίτερο σε περίπτωση παραπτώματος. Ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται διαχωρισμός και διάκριση εδώ. Όλοι οι οποίοι παραβιάζουν τον οδικό κώδικα θα πρέπει να ε, τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο. Όσον αφορά ε, το ενόπνευμα ε, και την οδήγηση ε, συμφωνώ ότι πρέπει να απαγορευτεί ο συνδυασμός αλλά πιστεύω ότι η τροπολογία Βιντάντσα δεν ε, αρμόζει στο σημείο αυτό. Επίσης όσον αφορά την αλλαγή εκπαιδεύσεως για μείωση των συγκρούσεων δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε εμείς να κάνουμε έχει σχέση με το θέμα μας εδώ η τροπολογία αυτή τεχνική παρακολούθηση των δικύκλων και των μοτοποδηλάτων ε, νομίζω δημιουργεί μία παρανόηση διότι εγώ αναφέρθηκα εις τα μοτοποδήλατα και τα δίκυκλα μετά από ένα ατύχημα και ε, κάθε όχημα το οποίο ε, μπλέκεται σε ε, ένα ατύχημα πρέπει να ελεγχθεί τεχνικά προτού να μπορέσει να κυκλοφορήσει πάλι. Επίσης ε, έχω και άλλα ερωτήματα αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ οι συντάκτες των τροπολογιών και έτσι δεν μπορούν να μου τα διευκρινίσουν. Η κυρία Γιάλα Σέντερ παραδείγματος χάρη ε, ε, αναφέρεται εις την ζημία του οδοστρώματος σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν το καταλαβαίνω, θα πρέπει να μου το εξηγήσει. Ε, ε, όσον αφορά μια άλλη τροπολογία θα ήθελα πληροφορίες για να δω πώς μπορούμε να το ενσωματώσουμε στο κείμενο. Η κυρία Σεναλόβα ε, ε, ε, ζητά να υπάρξει εκπαίδευση οδηγών ε, από όλα τα επαγγέλματα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί εδώ και θα ήθελα να μου το εξηγήσει. Υπάρχει και μία αίτηση του κυρίου Κούκλιας ο οποίος ζητά να υπάρξει μέχρι το 2023 ενιαίος κόξ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό σημαίνει ότι στη Μεγάλη Βρετανία θα αλλάξουν και αντί από δεξιά θα πηγαίνουν αριστερά ή αντιστρόφως. Κάποιος θα έπρεπε να μου το εξηγήσει αυτό. Ο κύριος Στέρξ παραδείγματος χάρη μας λέγει ότι χρειάζεται ε, μια καλύτερη παθητική ε, ε, επάνδρωση των δρόμων και όταν μιλάω για ευέλικτο φωτισμό των δρόμων θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι εννοείται. Επίσης ε, όσον αφορά το, την τροπολογία του κυρίου Σίμψον ε, για τους ε, ποδηλάτες ε, δεν αντιλαμβάνουμε τι εννοείται γιατί εγώ δεν ερμηνεύω με τον ίδιο τρόπο τη διατύπωση που χρησιμοποίησατε. Και τέλος άλλα θέματα όπως σας είπα θα συντονιστούν σε συμβιβασικές προτάσεις για τη διαβίου μάθηση, για την προστασία των δεδομένων ε, θα υπάρξει μία συμβιβαστική τροπολογία για τις ιατρικές εξετάσεις, επίσης ε, ε, για την πρακτική εφαρμογή της περαιτέρω εκπαιδεύσεως. Θα ήθελα να μου πείτε τι εννοείται με τα αλκοολόξ, με τα έξυπνα οδικά συστήματα, και τέλος όσον αφορά τον Ευρωπαίο Συντονιστή ο κύριος Ελκαντράου, ο κύριος Ρικίε, Γιάλα Ζέντερ Κομουτσάκος και άλλοι ε, ε, ζητούν να ε, υπάρξουν διευκρινήσεις τις οποίες θα προσπαθήσω. Δεν θέλω να υπάρξει ένας αυτόνομος οργανισμός αλλά θα ήθελα να υπάρχει αναγνωρισμένος κάποιος συντονιστής για την οδική ασφάλεια ο οποίος με τις εμπειρίες του θα μπορέσει να προωθήσει την έρευνα και την εφαρμογή ε, μιας ε, πολιτικής στο χώρο και να εναρμονίσει τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στα διάφορα κράτη όπως άλλωστε και τις πρακτικές για να μπορέσει να εφαρμοστεί καλύτερα το δίκαιο και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Όλες αυτές είναι προτάσεις που έχουν έχουν ε, υποβληθεί για να ε, καταρτήσω μία πιο συγκεκριμένη ε, έκθεση και θα προσπαθήσω εντός της εβδομάδας να καταλήξω σε ένα πιο ακριβές κείμενο το οποίο θα υποβάλουμε και στην Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα έχουμε αίσιο αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και πάλι έχουμε ένα πολύ μακρύ κατάλογο μιλητών. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Για τους σκιώδεις ηγητές θα δώσω τρία λεπτά στον καθένα, ενώ στους άλλους ομιλητές θα ζητήσω να μιλήσουν μέχρι στο δύο λεπτά, γιατί αλλιώς δεν θα μας περισσέψει χρόνος. Σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα αυτό αφορά τις τροπολογίες της ίδιας, παρακαλώ να μην επαναλάβουμε τα κεντρικά μας σχόλια. Κυρία Σεναλόβα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ε, σοσιαλιστή Σκιώδη εισηγητή, ομιλώ, ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προσπάθειες του. Έχει πολλές τροπολογίες μπροστά του, αλλά αυτό δείχνει και το σημαντικό ενδιαφέρον που εκφράζουν τα μέλη για το ζήτημα αυτό. Οι τροπολογίες ε, δεν είναι ένας ε, Δεν είναι μια προσβολή, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ήδη καλή δουλειά του εισηγητή. Ο εισηγητής ανακοίνωσε πολλές συμβαστικές προτάσεις Θα εστιαστώ σε μερικές από αυτές. Πρώτον, ο Ευρωπαίος συντονιστή οδικής ασφάλειας. Το θέμα αυτό είναι έτσι αμφιλεγόμενο. Εμείς υποστηρίζουμε αυτό το θεσμό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε ε, συνένεση στην εναρμόνιση των οδικών κανόνων προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Μετά, διπλώματα οδήγησης. Περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια, στην οδική ασφάλεια, ε, η λεπτομερής ανάλυση των ατυχημάτων, κάτι που απαιτεί η δεδομένη υψηλής ποιότητας, ασφαλείς υποδομές και μέτρα εναντίον της οδήγησης με την επίρρεια ναρκωτικών και ινοπνεύματος. Όλα αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα για τον δικό μας και δυσηγητή. Θα πρέπει να αναζητήσουμε λοιπόν μια λύση, μια συμβαστική λύση για αυτά. Σε ό,τι αφορά το οδήγηση υπό την επίρρεια υπομέθη, ε, να πω κάτι προσωπικό, ένα προσωπικό μου σχόλιο. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό όριο, μέγιστο όριο ε, για την περιεκτικότητα του αίματος σε ε, αλκοόλ. Πιστεύω το 0% που ήδη υπάρχει σε 6 χώρες θα ήταν το κατάλληλο όριο. Ευχαριστώ. Κρίσπεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Κόχ και όλους τους ε, συναδέλφους ε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά τους τελευταίους μήνες. 272 οι τροπολογίες, κάτι που δείχνει το ενδιαφέρον των συναδέλφων. Χωρίς να ε, επανέλθω σε αυτά που έχουμε ήδη πει, να σχολιάσω αυτές τις τροπολογίες που είναι πιο σημαντικές για μας και θα θέλαμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Οι συνάδελφοι ε, Γκούτσιας και Στέρκ έχουν ε, υποβάλει επίστηκες τροπολογίες. Θα επανέλθω την Πέμπτη για να απαντήσω και στις ερωτήσεις του Ντίτερ. Θα έρθω σε επαφή μαζί τους. Λοιπόν, το θέμα του συντονιστή, πολύ σημαντικό για μας. Δεν, μας, δεν θεωρούμε ότι είναι ε, απαραίτητη η δημιουργία αυτού του θεσμού. Πολύ συχνά στην ε, Ευρώπη δημιουργούμε θεσμούς που ε, δεν είναι σαφής η αποστολή τους, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να πάρουμε μία ακόμα τέτοια απόφαση. Αντιθέτως πιστεύω ότι θα προσθέταμε μεγαλύτερο άχθος στο σύστημα πιστεύω ότι θα ήταν καλό αυτές οι αρμοδιότητες να ε, υλοποιηθούν, να αναλυφθούν σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, για την κατάρτιση. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ε, έχω την εντύπωση πως προέκυψε η ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων κινητικότητας εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που ε, είναι ανάμεσα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την ΣΑΡ της ε, Γαλλίας, ε, στο, στην καρδιά μια ζώνη τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε πέρασμα λοιπόν, στα σταυροδρόμοι και γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε κοινό ορισμό για ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ε, για τους κινδύνους, ποια ακριβώ είναι η κίνδυνη, αν η κατάρτιση, ανεξαρτήτως του αν μιλούμε για ποδηλάτες, ε, μοτοποδηλάτες κλπ, ε, μοτοσυκλετιστές κλπ, οι τα διασυνοριακά πρόστιμα και ποινές, κυρώσεις, έχουν καταθεί πολλές τροπολογίες για αυτό το θέμα θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό ορισμό. Ε, χρήση συστημάτων ε, ε, εξουδετερώση των οχημάτων σε περιπτώσεις ε, ε, οδήγησης με την επίρρεια αλκοόλ. Υπάρχουν ήδη κανόνες για τους οδικούς φορτηγών που ε, προσπαθούν να οδηγήσουν ε, σε κατάσταση μέθησο και εδώ θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς. Ε, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, αλλά θα τα πούμε αυτή τη βδομάδα, την Πέμπτη. Ευχαριστώ. Thank you for that. Mr. Taylor, minutes. Ο Τέιλορ, τρία λεπτά, παρακαλώ. Ο Τέιλορ, τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ταχύτητα αλκοόλ και ναρκωτικά είναι κακό κοκτέιλ, επικίνδυνο κοκτέιλ και κατά της ασφάλειας. Δεν ε, πρόσεξα ότι αναφερθήκατε στην ταχύτητα στα εισαγωγικά σας σχόλια, αλλά σήμερα το πρωί στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ασφα... Οδικής Ασφάλειας ε, έμαθα ότι η ταχύτητα ευθύνεται για το 1 τρίτο όλων των ε, θανατηφόρων ατυχημάτων. Και για το λόγο αυτό θα συνιστούσα στα μέλη να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία της ε, τροπολογίας 126, δηλαδή να προαγάγει η Κομισιόν ένα όριο ζώνης 30 χιλιόμετρων σε κάποιες ε, περιοχές, ιδιαίτερα γύρω από σχολεία και σε κατοικημένες ζώνες στις ζώνες ε, κατοικίας. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να στοχεύσουμε σε ευαίσθητες περιοχές, θα πρέπει να στοχεύσουμε στα σχολεία, στην εκπαίδευση και θα πρέπει ε, να είναι υπέρ των συμφερόντων των πεζών, των ποδηλατών και θα πρέπει να εξασφαλίσει μια αποτελεσματικότερη επιβολή της υφτάμενης νομοθεσίας και των νόμων. Θα πρέπει να μετακινήσουμε το πρότυπο μακριά από τα γεωταχή, μακριά από τα αυτοκίνητα και υπέρ των επαγγελματικών οχημάτων. Άκουσα τα σχόλια του κυρίου Κόχο σχετικά με το εξωτερικό κόστος ε, που επιφέρουν τα ατυχήματα και ότι αυτό θα πρέπει να εσωτερικευθεί, με συγχωρείτε. Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη ζωή συχνά παρατηρούμε ε, τα πράγματα όσο περισσότερο κοστίζουν. Εάν αγνοήσουμε τις δαπάνες, τα έξοδα των ατυχημάτων, τότε αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε τα διδάγματα που θα έπρεπε να έχουμε από την επιβολή της ασφαλείας. Ευχαριστώ, πρόεδρε, λέει ο κύριος Bradburn. Κοιτώ τις τροπολογίες και κατανοώ γιατί δεν πιστεύω ότι η λύση στα θέματα της οδικής ασφάλειας είναι η περισσότερη Ευρώπη. Αλλά θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής, πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες με τις οποίες συμφωνώ, δηλαδή όλες αυτές που θα διαγράψουν την οποιαδήποτε αναφορά σε έναν Ευρωπαίο συντονιστή ε, για την οδική ασφάλεια. Αυτό ακριβώς είναι που δεν χρειαζόμαστε. Ο κύριος Κοχ ε, υπογράμμισε κάποιες προβληματικές περιοχές και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Το θέμα είναι ποιες είναι οι λύσεις. Αυτό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα. Τώρα οι, ανότι, οι ανόητες ιδέες εναρμόνισης των οδικών, της οδικής σήμανσης και όλα αυτά που έχουμε διαβάσει για τους ποδηλάτες, ελπίζω πραγματικά να συμφωνεί ο κύριος Κόχο ότι είναι πραγματικά ανόητα παραδείγματα. Τώρα, το πρόβλημα της ε, μέθης. Όπως είχα πει στην προηγούμενη συζήτηση, Πρόεδρε, και εδώ αναφέρουμε στροπολογίες που αναφέρονται σε αυτά τα όρια του αλκοόλ κτλ. Υπάρχουν περισσότερες λύσεις για ένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία συνέχεια. Στις περιπτώσεις που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπο... οι, ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποσύρονται γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το κόστος, το αυξανόμενο κόστος της κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων περιστατικών. Δεν χρειάζεται συνέχεια περισσότερη νομοθεσία για τις κυρώσεις ε, και το κλείδωμα των οχημάτων σε περίπτωση τέτοιων παραβιάσεων. Και αυτό μπορεί να οδηγούσε σε, μια, σε ένα περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά μετά θα έπρεπε να περάσουμε και στην, στο περιορισμό των, ε, της κατανάλωσης ε, ναρκωτικών Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ξαναπώ ότι υπάρχουν κάποιε καλέ ιδέε τη τροπολογία που πρέπει να ενθαρρυνθούν, αλλά δεν χρειάζεται όλα αυτά τα σημεία να καλύπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλούμε για την καθοδήγηση των παιδιών και την οδική ασφάλεια. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, όπω ξέρετε, Πρόεδρε, αυτό υπήρξε πάντα ε, υπό την αιγίδα τη σχολική εκπαίδευση από τι πρώτε βαθμίδε. Από τι πρώτε τάξει του σχολείου δεν χρειάζεται να έχει σχέση με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Οποιαδήποτε χώρα γνωρίζει ότι αυτά είναι αυτά που θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά ούτω ή άλλω. Δεν θα επιμηκύνω τη συζήτηση εδώ, Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι έχουμε καθυστέρηση, αλλά θα πω απλώ ότι το σκεπτικό είναι σωστό, αλλά οι πρακτικέ λεπτομέρειε είναι τελείω λανθασμένε κατά την άποψή μου και να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Κόχ πρέπει να αποχωρήσω πριν το τέλο τη συζήτηση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 Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόχ για την έκθεσή του που έχει φιλόδοξους στόχους για την βελτίωση της ε, οδικής ασφάλειας και αναφέρεται και στους ε, εποχούμενους και γι' αυτό χρειάζεται και νέες διατάσεις. Αναφέρεται συγχρόνως και στους πεζούς και στους ποδηλάτες και θα πρέπει ε, τα μέτρα υποδομής για τους πιο αδύναμους συμμετέχοντες στη συνοδική κυκλοφορία όπως η πεζή και οι ποδηλάτες να ενισχυθούν. Ε, η Άλντε στηρίζει, οι φιλελεύθεροι δηλαδή στηρίζουν την τροπολογία 16 ε, και ε, αποβλέπουν στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων στην οδική κυκλοφορία Ιδίω για πεζούς και ποδηλάτες και τη μείωση των ε, θανατηφόρων ε, ε, ατυχημάτων κατά 50%. Ε, θα έπρεπε να εξεταστεί ε, επίσης ε, συγκεκριμένα και αυτό γίνεται μέσω μιας τροπολογίας η όραση και επίσης θα ήθελα με την τροπολογία 126 να στηρίξω ότι 30% όριο ταχύτητος θα έπρεπε να υπάρχει στις πόλεις και 120 στον αυτοκινητόδρομο εκτός από τα δίκτυα ταχείας ε, κυκλοφορίας. Επίσης ε, θα θέλαμε να συμφωνήσουμε με την τροπολογία των ε, των ε, σοσιαλιστών για μία μείωση στο 0,2% ο κύριος Κόχο θα ήθελα ε, να υπερισχύσει όσον αφορά το τυφλό σημείο της οπτικής γωνίας των φορτηγών και γενικώ τον συγχαίρω για την έκθεση. Ευχαριστώ εάν ο τελευταίος, οι τελευταίοι ομιλητές μπορούν να περιοριστούν σε δύο λεπτά θα μπορέσουμε να καλύψουμε το χρόνο. Ο κύριος Κράμερ, κύριε Κόχο, δεν τα σκεφτήκατε όλα διότι 50% των ατυχημάτων ε, οφείλονται εις το, ε, εις το ενόπνευμα ή εις την κόποση και γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε στο 0,2% και είχαμε ένα τεράστιο ατύχημα στην Γερμανία θανατηφόρο οπότε γιατί ε, να υπάρχουν αυξήσεις του ορίου ταχύτητας και να μην μείνουμε στα 80 χιλιόμετρα. Επίσης, ε, όσον αφορά τη, τα κράνη που έπρεπε ε, να τα ε, φορούν πέραν των δικύκλων και οι οδηγοί στα αυτοκίνητα, στον αυτοκινητόδρομο, δεν συμφωνώ. Δεν πρέπει να περιπλέκουμε την κατάσταση στους αυτοκινητοδρόμους όμως γιατί ε, στο Άμστερνταμ ε, ε, φορούν, δεν φορούν ειδικό σακά, γυλαίκο και ειδικό ο κράνος για να μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη και εκεί ίσως θα πρέπει να επιτείνουμε τους, τα όρια ταχύτητος και την προσοχή ε, και να μην περιπλέκουμε την κατάσταση. Τέλος, ε, κάνατε είδατε μία εκδήλωση ε, του λόμπι αυτών που κατασκευάζουν αυτά τα γυλαίκα το οποίο όμως δεν καθορίζει ούτε επηρεάζει την πολιτική ασφαλεία των οδικών μεταφορών. Ε, κύριος Ρικέ. Θα ήθελα να πω το εξής. Ένα πράγμα, λεπτομέρεια βέβαια, αλλά σημαντικό. Στην προβληματική των ναρκωτικών και του αλκοόλ, ο κ. Σόσμπαντ είπε ε, μίλησε για τους ε, πόντους που χάνονται, τους βαθμούς που χάνονται από το δίπλωμα. Αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό αυτό το σύστημα. Πρέπει να διαθέτουμε ένα σύστημα αυτόματου κλειδώματος που θα εμποδίζει να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας όταν κάποιος είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ε, ναρκωτικών βέβαια με δικά του, δικές τους δεν θα είναι, δεν πρέπει η κοινωνία ή η ε, βιομηχανία να το πληρώσει. Αντί να χτυπάει καμπανάκι όταν δεν βάζει κάποιο στη ζώνη του, α βάλουμε αυτό το σύστημα που θα κλειδώνει την ε, μηχανή και έτσι θα γλιτώνουμε το 50% των ατυχημάτων. Δεν είναι και τόσο ε, μάλιστα ακριβό, οπότε δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Minutes, Κυρία Μάης, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζομαι καν δύο λεφτά, διότι ήθελα να συμπληρώσω αυτό που δεν πρόλαβε να πει η κυρία Γκρίσμπερκ σαν όδηση συγγήτρια, δηλαδή τα μέτρα ασφαλείας για τους ποδηλάτες και για άτομα που χρήζουν βοηθείας, επίσης εναρμόνιση για τα μιλιχιλιοστά που χρειάζονται στην κατανάλωση ε, νοπνεύματος και ε, Επίσης ε, πιστεύω ότι πρέπει να ρυθμίσουμε και τους περιορισμούς της ταχύτητας. Ε, ε, όσον αφορά τον κύριο Στέρξ ε, και ε, την ε, τον ευέλικτο φωτισμό προέρχεται από το Βέλγιο που φωτίζουν πολύ περισσότερο τους δρόμους από τη Γερμανία και ίσως πρέπει να δούμε όχι αν έχει οδηγήσει πάρα πολύ χρόνο ο οδηγός αλλά τι χρειαζόταν. Με συγχωρείτε διότι Νομίζω ότι σας έδωσα 30 ε, δευτερόλεπτα λιγότερο από ό,τι έπρεπε, ε, κυρία Γκρίσμπεκ, και σας ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Μάισνερ όμως σας συμπλήρωσε. Ο κύριος Μπακ για δύο λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, γενικά θα ήθελα να συμφωνήσω με τις εκτιμήσεις του κυρίου Κοχ και οι πολλές από τις τροπολογίες αναφέρονται εις ε, την, ε, τις υποδομές ε, του οδικού συστήματος τις οποίες χαιρετίζουμε, χρειάζονται αλλά και γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρεί ότι πρέπει να μειώσουμε τις, την κυκλοφορία ατομική ηλεκτρικών οχημάτων και μεγαλύτερη χρήση των ε, ε, μέσων, ε, δημοσίων μέσων μεταφοράς. Όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει, θεωρώ ότι είναι σημαντική και θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί στο πρόγραμμα. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι έχει σχέση με την εκπαίδευση και όσον αφορά την παρακολούθηση διασυνοριακά για παραπτώματα και ευαισθητοποίηση νομίζω ότι καλό θα ήταν να συνεργαστούμε εις τον τομέα της οδικής κυκλοφορίας και όσον αφορά το, την τροπολογία 30 ε, πιστεύω ότι μία παγκόσμια ημέρα κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντική ε, και ε, υιοθετείται από το ΝΟΙΕ και από την Διεθνή Οργάνωση Υγείας για να μπορέσει να τονίσει και την τραγωδία των ατυχημάτων και να ευαισθητοποιήσει το κοινό. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένας, μια παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησεως. Ο κ. Δεγκράντες. Να πω καταρχήν ότι η έκθεση Κόχ είναι εξαιρετική. Και δεν είναι τυπικό αυτό που λέω, το εννοώ. Ε, φυσικό όμως να υποβληθούν πολλές τροπολογίες. Ε, όλοι νομίζουν ότι γνωρίζουν το ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι εύκολο κανείς να σχολιάσει, οπότε είναι φυσιολογικό να υφίστανται τόσε τροπολογίε. Ο εισηγητή θα δυσκολευτεί βέβαια να ξεχωρίσει ποιε από αυτέ πρέπει να ικανοποιηθούν. Εγώ υπέβαλα δύο τροπολογίε που ενδεχομένω δεν εμπίπτουν ε, βέβαια σε όλο αυτό το όμνιμπους στο, στο οποίο, το οποίο συζητάμε. Ε, το θέλω να σχολιάσω τις στατιστικές. Ε, πρώτον, η, η ξεκούραση, η ανάπαυση του σημείου 28. Θέλω να πω το εξή. Τώρα που έχουμε τον ψηφιακό ταχογράφο και είναι δυνατόν οι οδηγοί μεγάλων αποστάσεων να μπορούν να επιστρέψουν αντι, ε, ε, μπορούν να επιστρέψουν, ε, ε, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί αυτή η διάταξη, γιατί η απουσία αναπαύσεων δημιουργεί ατυχήματα. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μεγάλα φορτηγά τα οποία από μόνα τους μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά ατυχήματα. Δεύτερον, να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις υποδομές τους εκεί ιδιαίτερως όπου εντοπίζονται ε, ιδιαίτερα προβλήματα με αυξηλούς ε, δείκτες ατυχημάτων. Χρειάζεται να λαμβάνονται μέτρα διόρθωση, διορθωτικά μέτρα, όχι οπουδήποτε, όχι σε όλα τα σημεία του δικτύου, αλλά εκεί που εντοπίζονται μεγάλοι ψηλοί δείκτες ατυχημάτων. Τέλος, πω το εξή. κάναμε, ε, κάποια στιγμή αντί για αυτοκινητοδρόμους είχαμε αποφασίσει στην Ισπανία να φτιάχνουμε, να διαπλατείνουμε τους παλιούς δρόμους, μικρού δρόμου μας. Ε, χωρίς ε, διαχωριστικό διάζωμα στη μέση. Αυτό δημιουργεί σημαντικότατα προβλήματα. Είναι δύσκολο να διορθωθεί, αλλά πρέπει να διορθωθεί. Ευχαριστώ. you, Sender. minutes, please. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Δύο λεπτά. Και εγώ συγχαίρω τον κύριο Κόχ. Έχει πολύ τεχνογνωσία, γίνει πολύ οργανωτικός, γνωρίζει και το θέμα πολύ βαθιά. Νομίζω ότι η έκθεση ήταν εξαιρετική. Οι τροπολογίες ε, έχουν ως μόνο στόχο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το ε, σύστημα που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τα ατυχήματα. Ε, οι δικές μου τροπολογίες έχουν σχέση με το σύστημα των υποδομών. Με συγκεκριμένες προτάσεις για το σχεδιασμό, ε, για τις ε, πληροφορικές πινακίδες και όλα αυτά, όλο, όλο, όλο αυτό το φάσμα και δεν μιλάμε μόνο δηλαδή για την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων αλλά και όλα όσα την ακολουθούν και τη συνοδεύουν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της οδικής ασφάλειας. Δεύτερον, οι ευάλωτοι χρήστε, για παράδειγμα μοτοσυκλετιστέ και δικυκλιστέ γενικότερα. Εκεί έχουν μειωθεί λιγότερο τα ατυχήματα από ό,τι στου άλλου και θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο αυτήν την ομάδα χρηστών. Ε, ευχαριστώ πολύ για την 120 ε, ε, για την πρόσκληση που μου απευθύνθηκε να υποβάλω την 120. Ε, Επίσης για τους ε, μετακινούς εργαζόμενους ε, είναι πολύ σημαντικό να εστιαστούμε και σε αυτούς γιατί γίνονται όλο και πιο μεγάλη ομάδα. Και μετά βλέπω ότι υπάρχουν όλο και, περισσότερες, ε, και περισσότερη υποστήριξη για την εναρμόνιση του ε, ανώτατου ορίου ταχύτητας και της ε, περιεκτικότητας του ανώτατης περιεκτικότητας αίματος σε αλκοόλ. Ε, αυτό το 0% που προτάθηκε και που ισχύει σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντσάν, δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον ε, συνέλφο Κόχο για τη δουλειά. Νομίζω ότι έχουμε αρκετέ προτάσει δυνατότητά μα ε, και στη δυνατότητά του ώστε να, να τις χρησιμοποιήσει κατά τον πιο κατάλληλο τρόπο για υπέρ της οδικής ασφάλειας στους δρόμους μας. Ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Οι ε. χώροι στάθμευση, καταλήλω εξοπλισμένοι κατά μήκος των εθνικών οδών, είναι ένα σημαντικό στοιχείο Σήμερα αυτό δεν ε, το παρακολουθούμε επαρκώς, ούτε το εξασφαλίζομαι. Αυτοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία κατά μήκο των δρόμων, ώστε και οι μεταφορείς, οι οδηγοί κτλ. θα πρέπει να μπορούν να τους χρησιμοποιούν κοντά και σε πρατήρια βενζίνης και και ανεφοδιασμού. Νομίζω ότι αυτό καλό θα ήταν να εισαχθεί μέσα στο σχεδιασμό γιατί είναι σημαντικό ζήτημα πιστεύω για την ασφάλεια των εθνικών οδών. Θα έπρεπε να προσέξουμε και περισσότερο την τροπολογία την 99 που αφορά την εξοικονόμηση αλλά αφορά και την θέση οδήγησης η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ηρεμία αν θέλετε και τελικά την ασφάλεια του οδηγού. Αυτά εντός των δύο λεπτών που είχα στη θέση μου πρόεδρε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ ο κύριος Higgins δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέντε σύντομα σημεία. Καταρχά, συμφωνώ απολύτως για τι τροπολογίε 10 και 11. Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα προκύπτουν σε δευτερεύουσες οδούς και όχι στις βασικές εθνικές οδούς. Τώρα, έχουμε σε σχέση με, με το θέμα της ασφαλούς οδήγησης ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο και κάτι απολύτως κρίσιμο. Η τροπολογία 93. Το οπτικό πεδίο είναι πολύ σημαντικό για την ικανότητα οδήγησης και εκεί έχουμε μεγάλη ασάφεια και απόκληση στο τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα ελάχιστο, μια δοκιμή ελάχιστου οπτικού πεδίου και όρασης αν δούμε στο Βέλγιο δεν υπάρχει καθόλου τέτοια δοκιμή. Στη Γαλλία θα πρέπει να αποδεικνύει κανείς ότι έχει ένα πρόβλημα. Στην Φιλανδία και στην Ιλλανδία έχουν... πρέπει να αποδεικνύει και πάλι κανείς ότι η όρασή του είναι στο κατάλληλο πεδίο. Επίπεδο, με συγχωρείτε. Αυτό που αποκαλούμε τρίφτες Πρόεδρε. Είναι πολύ φθηνή, αλλά είναι πολύ κίνδυνη. Στην ουσία έχουμε ένα όριο μεταξύ των δύο, ε, ε, των δύο κατευθύνσεων κίνησης των οδών, οι οποίες πολλές φορές είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα, τα αν θέλετε, κυκλειδώματα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρο ατύχημα. Αυτό αποκαλούμε τρίφτες ε, στα αγγλικά. Cheese graces, είπε ο μιλητής. Το 2033 μόνο τότε θα έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης και τότε ίσως θα μπορέσουμε να αρμονίσουμε αυτά τα στοιχεία. Πρόεδρος, καταρχάς, έχοντας ακούσει τα όσα είπε και ο κύριος ε, Higgins, ο κύριος Κοχ είχε ερωτήσει σχετικά με τα κυκλειδώματα αυτά προστασία. Ένα από τα προβλήματα που σχετίζεται με αυτό, με τα μεταλλικά πολλές φορές είναι πράγματι πολύ επικίνδυνα αλλά πολύ συχνά προεξέχουν διάφορες βίδες και στοιχεία των κυκλειδωμάτων και πολύ συχνά αυτά ακριβώς προκαλούν θανατηφόρα ατύχημα, ατυχήματα, ειδικά για τους μοτοσυκλετιστές. Αυτά τα μεταλλικά κυκλειδώματα αυτή τη στιγμή επίσης δεν σταματούν οχήματα αρκετά βαριά να περάσουν από την αντίθετη κατεύθυνση όταν υπάρχει ατύχηματα. Ενώ τα τυχεία για παράδειγμα από σκυρόδεμα, έχουν πιο όλια επιφάνεια και σταματούν το όχημα. Και πολύ συχνά έχουμε την ε, δυνατότητα να αποφύγουμε το θανατηφόρο ατύχημα γιατί ακριβώς η επιφάνεια είναι ομαλή και λία και δεν έχει όλες αυτές τις υπερεξοχές που έχουν τα μεταλλικά κυκλειδώματα. Το άλλο που ήθελα να πω άκουσα για τις ε, αναπαυτικές ε, θέσεις οδήγησης και για τα για τα ταξί. Πολύ συχνά είναι τόσο αναπαυτικές οι θέσεις που ενθαρρύνουν κάποιον να αποκοιμηθεί, είχε πει κάποιος. Εν πάση περιπτώσει είναι κρίμα που έφυγε ο κύριος Bradburn γιατί όταν μας είπε για τον έλεγχο ε, των ορίων αλκοόλ και τις ασφαλιστικές ε, ε καλύψεις που είναι τόσο Ακριβέ, Ένα από τα προβλήματα έχει στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή είναι ο αριθμό των ανθρώπων που κυκλοφορούν χωρί ασφάλιση γιατί δεν μπορούν να την πληρώσουν. Και αυτό σημαίνει ότι σταματούν να οδηγούν. Όχι. Κυκλοφορούν στον δρόμο χωρί να είναι ασφαλισμένοι. Επομένω το επιχείρημα, και νομίζω και ο Ντομινίκ ε, το, το ανέφερε, ε, είναι απολύτω ανόητο. Εκεί χρειάζεται επιβολή αποτελεσματική των ορίων. Τώρα, πολύ γρήγορα. Ξέρω, κύριε Πασκουαρέλη, ότι έχει αυξηθεί η πίεση προ την περιοχή σας όλη την, ε, τη διάρκεια όλης της αλλά έχετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε τα τελευταία και να κλείσουμε στο 12.30. Ευχαριστώ. Το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα λεπτό γιατί οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες είναι κατακαιρματισμένες, ελάχιστες υπάρχει θέμα επικουρικότητας το οποίο επικαλούνται πολλά και δικαίως πολλά κρατημέλη και ταυτόχρονα υπάρχει μια ισχυριότατη ζήτηση από τους, ε, πελάτες, από τους ε, πολίτες μας. Η Ευρώπη έχει λοιπόν ρόλο να παίξει, είναι αποτελεσματικός ρόλος, ε, χωρίς υπερβολική εναρμόνιση, χωρίς πολυγραφειοκρατία. Ο κύριος Κόχ στην έκθεση του αναφέρει. Ο αριθμός των τροπολογιών πολύ υψηλός αποδεικνύει άλλωστε την, αυτή την υψηλή ζήτηση, πληρία ανάγκη να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως Ευρώπη σε ένα θέμα το οποίο αγγίζει την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών μας. Προφανώς δεν πρόκειται να σχολιάσω τις διάφορες τροπολογίες. Ε, έχω όμως να κάνω ορισμένα σχόλια για συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το συντονιστή οδικής ασφάλειας. Είναι μια καλή ιδέα πρέπει να αναλυθεί και πιο, είναι πιο ρεαλιστική από την ε, εναλλακτική δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας. Ο συντονιστής δεν πρέπει ε, να θεωρηθεί ως ε, ένα πρόσθετο στοιχείο γραφειοκρατίας, αλλά ο συντονιστής αυτός θα αποτελέσει ένα πρεσβευτή οδικής ασφάλειας που θα μπορέσει να κινητοποιήσει όλο το, ε, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την, ε, και να συντονίσει την δράση των κρατών μελών. Μετά γίνεται λόγος για την ενοποιημένη προσέγγιση, την κατανοημένη ευθύνη την, την ευθύνη που συμμεριζόμαστε όλοι μάλλον. Υπάρχει και μια ηθική διάσταση σε αυτό. Η, το, το ιδανικό μηδέν, το, δηλαδή ε, με, ε, μηδενικά ατυχήματα, ε, το βλέπουμε αυτό και στις ε, βόρειες και στη Λευκή Βιβλίο της Κομισιόν. Αυτό το όραμα μηδέν ε, δεν θα πρέπει να συγχαίεται με τους ποσοτικούς στόχους που έχουμε καθορίσει ναι, ε, να μειώσουμε κατά 50% τα, τους θανάτους μεταξύ του 2010 και 2020, όπως το είχαμε κάνει και μεταξύ του 2000 2010. Ε, το όραμα 0 δεν είναι ένας ποσοτικός στόχος, είναι μια φιλοσοφία ε, που, ότι, που βασίζεται στην θεώρηση ότι δεν επιτρέπεται άνθρωποι να πεθαίνουν στον δρόμο. Στο πλαίσιο αυτού του οράματος χρειαζόμαστε και ποσοτικούς ποσοτικοποιημένους στόχους. Μείον 50% τα επόμενα 10 χρόνια λοιπόν. Αυτό θέλουμε να το διατρήσουμε ως γενικό στόχο. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να καθορίσουμε ενιαίους στόχους ανά κατηγορία χρηστών, για παράδειγμα ηλικιωμένοι παιδιά, ε, πεζή. Ε, και κλπ. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε και προβλήματα ε, υπολογισμών, θα ήταν και μακάβριο και ταυτόχρονα θα αύξανε και τη γραφειοκρατία. Ένα στόχος είναι πολιτικά ισχυρό μήνυμα. Και όταν μιλάμε για πολιτικοποιημένους στόχους θα πρέπει να βελτιώσουμε τα στατιστικά εργαλεία που διαθέτουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μιλάμε για το δίπλωμα οδήγηση. Οι μελέτε που αυτή τη στιγμή διεξάγει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των, των συστημάτων ε, βαθμολόγηση, ε, ποινών με βαθμού, ε, δείχνουν ότι ότι το ενοποιημένο σύστημα διπλωμάτων θα τεθεί σε, σε ισχύ από το 2013 και όχι το 2013 και μετά. Ε, μετά έχουμε το θέμα των κυρώσεων, διαδικτυακών κυρώσεων, έχουμε το θέμα των υποδομών. Τις υποδομές θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε στους χρήστες σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Ευρώπη των 27 θέλουμε να εναρμονίσουμε τις πινακίδες. Υπάρχουν διεθνείς ε, συμβάσεις έτσι και αλλιώς που καλύπτουν μια γεωγραφική περιοχή πολύ πιο πλατιά από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εθνικές, ε, ε, εθνικοί κανόνες. Τέλος, ανακοινώνω μια νομοθετική πρόταση κομισιών που θα υποβληθεί στο μέλλον για την αναθεώρηση των κανόνων περί τεχνικού ελέγχου ε, οχημάτων και μια εμβάθυνση της στρατηγικής σε ό,τι αφορά τους ευάλωτους χρήστες και τους τραυματίες. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ. Ε, καταλαβαίνω ότι για ορισμένους η έκθεση είναι υπερβολικά προοδευτική, για άλλους όχι αρκετά, αλλά όσον αφορά το ενόπνευμα, ενιαία ρύθμιση για τα όρια σε όλη την Ευρώπη, για την πολιτική εσωτερικής αγοράς και υγεία συμφωνώ. Χρειαστεί όμως ένας συντονιστής για να συντονίζει τους διόφορους τομείς. Συμφωνώ ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους πολίτες και θα μπορούσε μπορούσε κανείς να μιλήσει με ψυχολόγους και εμπειρογνώμονες της κυκλοφορίας και να αποκομίσουμε συμπεράσματα. Επίσης στο Ροστόκο ε, είδατε ότι η μείωση της κυκλοφορίας δεν εμπόδισε το ατύχημα που οφειλόταν σε ένα ε, ε, άνεμο από άμμο και τέλος καλό έχει κανείς φανείς ε, οδηγίες όσον αφορά τις ιατρικές επισκέψεις νομίζω ότι θα συνεννοηθούμε ε, και όπως σας είπα θα κάνω συμβιβαστικές τροπολογίες και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά με τους ε, ε, σκιώδεις εισηγητές και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα έχετε καταλήξει όταν θα φτάσουμε στην ψηφοφορία η οποία στην Επιτροπή Μεταφορών προβλέπει Βλέπετε το Μάιο και στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Άρα Μάιος για την Επιτροπή, ο Ιούνιος για την Ολομέλεια και πριν χωρίσουμε για το μεσημεριανό η έκθεση Αγιάλα που θα είναι η πρώτη που θα εξετάσουμε σήμερα το απόγευμα στο 3 αναφέρεται ε, σε, στις ε, ε, μεταφορές ε, και διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας και υπάρχει σε όλες τις γλώσσες στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ, ξέρω ότι σας πίεσα, ε, να με συγχωρήσουν οι διερμηνείς που ξεπεράσαμε λίγο το όριο και θα σας δω όλους εδώ πάλι στις 3 ώρες.